Okay, friends. Uh, we start the second part of our... Αγαπητοί φίλοι, ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της σημερινής μας ε, συνεδρίασης και σας καλωσορίζω. Καλωσορίζω όλους τους συμμετέχοντες και φυσικά και τους ευρωβουλευτές. Σήμερα το πρωί είχαμε συζήτηση σχετικά με την ψηφιοποίηση για το πώς αλλάζει τις κοινωνίες μας, τη ζωή μας και τις αγορές εργασίας. Τώρα θα συζητήσουμε το ίδιο πράγμα σχεδόν. Θα μιλήσουμε για την παγκοσμιοποίηση, για τις θέσεις απασχόλησης που μεταφέρθηκαν σε άλλα μέρη του κόσμου και η ακρόασή μας έχει να κάνει με τον επαναπατρισμό των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Θα δώσω πρώτα τον λόγο στον κύριο Ρέιμον Τόρες, Διευθυντή του Τμήματος Ερευνών ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Και έχετε 10 με 12 λεπτά χρόνο ομιλίας. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό απόγευμα. Είναι προνόμιο να βρίσκομαι εδώ σήμερα να συζητήσω αυτό το θέμα σήμερα μαζί σας, το οποίο είναι σχετικά νέο και για το οποίο δεν έχουμε πολλά στοιχεία μέχρι στιγμής. Από πολιτικής πλευράς όμως είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα λοιπόν στην παρουσίαση να τονίσω κάποιες από τις βασικές τάσεις που σχετίζονται με τον επαναπατρισμό των θέσεων εργασίας και να συζητήσω κάποιους από τους παράγοντες και τις πολιτικές συνέπειες των τάσεων αυτών. Γνωρίζουμε ότι το reshoring, ο επαναπατρισμός ε, των θέσεων εργασίας είναι επιστροφή το κάποιων δραστηριοτήτων στην χώρα προέλευσης. Μεταφορά δηλαδή στην χώρα προέλευσης. Έχουμε στα αγγλικά τους όρους reshoring και backshoring, καθώς και nearshoring. Έχουμε κάποια σημαντικά παραδείγματα. Η Nestlé έχει μεταφέρει κάποιες από τις δραστηριότητε της από την Αφρική στην Ευρώπη και έχουμε και κάποιες σημαντικές τάσεις στις Ηνωμένε Πολιτείε. Βλέπουμε δηλαδή το φαινόμενο αυτό όχι μόνο στην Ευρώπη. Υπάρχουν παραδείγματα από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Όπως είπα και πριν, δεν είναι πολύ εύκολο να εντοπίσει κανείς τις τάσεις αυτές. Θα συγκεντρώσω λοιπόν όλες τις ε, πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Ξεκινάμε λοιπόν από την αύξηση στην ε, αναλογία σε σχέση με το ΑΕΠ καθώς ε, και το, την αναλογία ε, έτοιμων προϊόντων με τα ενδιάμεσα προϊόντα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι αυτή η μείωση στην αναλογία δείχνει ότι όλο και περισσότερα προϊόντα παράγονται εντός της Ευρώπης. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτός είναι ένας ε, δείκτης ο οποίος ε, συνάδει με, την, ε, με τον επαναπατρισμό παρότι δεν είναι απόλυτη απόδειξη για το θέμα αυτό. Κατόπιν έχουμε τον αριθμό των ανθρώπων που συνδέονται με τις αλυσίδες αξίας που υπάρχουν στον κόσμο αυτών, global value chains έχουν να κάνουν με τον κατακαιρματισμό των διαδικασιών παραγωγής ε, που βλέπουμε και εντός κάποιων χωρών ε, και ε, διασυνοριακά. Βλέπετε λοιπόν την γαλάζια γραμμή όπου βλέπουμε πτώση, δηλαδή οι άνθρωποι που εργάζονται εδώ φαίνεται να μειώνονται. Βλέπουμε δηλαδή σταθεροποίηση και μάλλον μείωση των ανθρώπων ε, που εργάζονται στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Και αυτό θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη ότι κάποιες ε, διαδικασίες που είχαν ανατεθεί εξωτερικά σε άλλες χώρες ε, τώρα συνεχίζουν να είναι αντικείμενο εξωτερικής ανάθεσης αλλά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλος σημαντικός δείκτης συνδέεται με τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Και εδώ βλέπουμε ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 και μέχρι και το 2005 είχαμε αύξηση, ενώ τώρα έχουμε μάλλον σταθεροποίηση και μικρή μείωση όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Και ενδιαφέρον είναι ότι για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια οι άμεσες ξένες επενδύσεις εντός της Ευρώπης που επιστρέφουν στην Ευρώπη είναι περισσότερες από ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις που ρέουν εκτός Ευρώπης. Για πρώτη φορά λοιπόν το 2012 που είναι τα τελευταία, τα πιο πρόσφατα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, Βλέπουμε περισσότερες επενδύσεις εντός Ευρώπης παρά Και αυτό δεν αποτελεί οριστική απόδειξη, αλλά ε, φαίνεται ότι αποτελεί ένδειξη για κάποιον επαναπατρισμό. Ε, βέβαια μπορεί να μην είναι επαναπατρισμός, μπορεί να είναι νέες δραστηριότητες, αλλά θα μπορούσε να οφείλεται εν μέρη στον επαναπατρισμό κάποιων θέσεων εργασία. Και το τελευταίο στοιχείο που έχουμε είναι ότι εξετάσαμε μία βάση δεδομένων που λέγεται FactSet που περιέχει εκατομμύρια μεγάλων επιχειρήσεων και διαπιστώνουμε και εδώ ότι το ποσοστό εγχώριων περιουσιακών στοιχείων φαίνεται να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Πραγματοποιείται δηλαδή όλο και μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής εντός της παραγωγής. Και αυτό μάλλον είναι πιο αξιόπιστος δείκτης ε, όσον αφορά τον επαναπατρισμό των θέσεων εργασίας. Ε, βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει κάποια αύξηση ε, στα περιουσιακά στοιχεία ε, των εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων. Επαναλαμβάνω όμως ότι και αυτό δεν αποτελεί οριστική απόδειξη ότι έχουμε μία μόνιμη και μαζική τάση επαναπατρισμού. Τα δεδομένα που έχουμε όμως ε, επιβεβαιώνουν κάποιες μακροοικονομικές μελέτες και διαπιστώσεις από με μεμονωμένες επιχειρήσεις. Οι μακροοικονομικές τάσεις λοιπόν επιβεβαιώνουν ε, αυτές τις ε, ενδείξεις που έχουμε εδώ. Βλέπετε στα τελευταία χρόνια την αύξηση των ε, εγχωριών περιουσιακών στοιχείων, όπως είπα πριν. Τα δεδομένα από τις μακροοικονομικές μελέτες δείχνουν ότι ο επαναπατρισμός περιορίζεται σε κάποιους τομείς. φαίνεται να πραγματοποιείται κυρίως σε τομείς όπου χρειάζεται πολύ κεφάλαιο και όχι πολύ εργασία, καθώς και ε, εκεί όπου χρειάζεται σημαντική εξειδίκευση των ε, εργαζομένων. Δεν βλέπουμε δηλαδή η μαζική επιστροφή των θέσεων εργασίας που μεταφέρθηκαν στην Κίνα. Μιλάμε για μεταφορά δραστηριοτήτων σε κάποιους ε, συγκεκριμένους τομείς. και μάλλον οι μεγάλες παρά οι μικρές επιχειρήσεις ε, φαίνεται να περνούν αυτή τη διαδικασία. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις ε, μακροοικονομικές μελέτες. Το βασικό ερώτημα είναι δεδομένου ότι έχουμε ε, ενδείξεις ότι γίνεται παραταπατισμός των θέσεων εργασίας. Για μένα το βασικό ερώτημα είναι γιατί γίνεται αυτό. Τρεις πιθανοί παράγοντες υπάρχουν. Ο ένας είναι ότι η, διαφορά στο κόστος ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες όπως είναι η Κίνα φαίνεται να μειώνεται κάπως. Δηλαδή, όσον αφορά την ε, περίπτωση της Κίνας, ε, υπάρχει αύξηση των μισθών 15 ε, έως 20% ανάμεσα στο 2000 και 2010. Έτσι μειώνεται η διαφορά στο κόστος, το οποίο σημαίνει ότι η Ευρώπη μπορεί να γίνεται πιο ανταγωνιστική. Και επίσης μπορεί να μειώνεται η διαφορά στο κόστος που συνδέεται με την αύξηση των, του κόστους μεταφορών λόγω της αύξησης των ε, τιμών των καυσίμων και άλλων ε, ε, δαπανών που συνδέονται με τις μεταφορές. Έτσι η παραγωγή κοντά στην κατανάλωση έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με πριν. Αυτό δηλαδή συνδέεται με το κόστος μεταφοράς και το κόστος των καυσίμων. Μπορεί λοιπόν και αυτό να αποτελεί έναν, παράγοντο, έναν παράγοντα που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ευρώπη ακόμα και σήμερα παρόλε τις εξελίξεις έχει μια σημαντική σταθερή δυναμική μέση τάξη με αγοραστική δύναμη, αυτό αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις επιχειρήσεις όταν ε, ε, σκέφτονται την μετεκατάσταση. Το δεύτερο θέμα είναι μάλλον πιο θεμελιώδες και σχετίζεται με τις νέες τεχνολογίες. Οι νέες τεχνολογίες όλο και περισσότερο καθιστά σημαντικό η παραγωγή να πραγματοποιείται κοντά στον καταναλωτή ώστε να υπάρχει άμεση αντίδραση στις αλλαγές στα ε, μοντέλα κατανάλωσης. Άλλος παράγοντας είναι η σημασία του να βρίσκεται κανείς κοντά στους χώρους όπου δημιουργείται η νέα τεχνολογία και η νέα γνώση. Κάποιες επιχειρήσεις λοιπόν που είχαν μετακατασταθεί επιστρέφουν διότι καταλαβαίνουν ιδιαίτερα σε τομείς έντασης κεφαλαίου και οπικές δεξιότητες όπου απαιτείται υψηλή εξειδίκευση, ε, μετεγκαθίστανται τώρα για να βρίσκονται πιο κοντά ε, ε, στα μέρη όπου παράγεται η νέα τεχνολογία και η ε, νέα γνώση. Ο τρίτος παράγοντας έχει να κάνει με τις κοινωνικές πτυχές. Νομίζω ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση, ειδικά στην Ευρώπη, αλλά γενικά, ότι η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με βάση κάποια πρότυπα εργασιακά, ε, κοινωνικά αλλά και περιβαλλοντικά και γι' αυτό υπάρχει ανησυχία για τα θέματα αυτά, ευαισθητοποίηση που μπορεί να οδηγήσει σε μετεγκατάσταση. Αυτό είναι άλλου τύπου επιχείρημα, το οποίο όμως έχει συνέπειες ως προς την πολιτική. Όσον αφορά την πολιτική, λοιπόν, θα πρέπει καταρχά να εξετάσουμε αν ο παναπατρισμό είναι κάτι θετικό ή αρνητικό. Βέβαια, αν επιστρέψουν θέσει απασχόληση στην Ευρώπη, αυτό είναι θετικό. Και ιδιαίτερα εάν πρόκειται για ε, θέσει απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων, ε, υψηλή τεχνολογία, υψηλής εξειδίκευσης. Ε, κάποιοι άλλοι παράγοντες όμως μπορεί να μην είναι τόσο θετική αν ε, συνδέονται με την ε, διάβρωση στην ε, ανάπτυξη κάποιων αναπτυσσόμενων χωρών. Για παράδειγμα, βλέπετε ότι στην Κίνα η κατάσταση δεν είναι τόσο καλή όσο ήταν πριν, οπότε μπορεί κάποιες επιχειρήσεις να μετεγκατασταθούν στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν θα υπάρχουν και τόσο πολλές εξαγωγές προς την Κίνα όσο υπήρχαν πριν. Ε, θα πρέπει να φροντίσουμε οι ε, αναπτυσσόμενες χώρες ε, να έχουν ροή κεφαλαίων. Υπάρχουν λοιπόν σίγουρα πολλά θετικά που συνδέεται με τον επαναπατρισμό των θέσεων απασχόλησης, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την προοπτική των αναπτυσσόμενων χωρών και θα πρέπει να διατηρήσουμε ένα δυναμικό κλίμα, να διατηρήσουμε μια σταθερή μεσαία τάξη και να στηρίξουμε τον κοινωνικό διάλογο στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Θα ήθελα να αναφέρω τρία είδη πολιτικών συνεπειών θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ελκυστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αποτελεί στόχο του επαναπατρισμού των θέσεων, της μετακατάστασης των θέσεων εργασίας. Κάθε χώρα μπορεί να κάνει πολλά για να βελτιώσει αυτή την ελκυστικότητα, να βελτιώσει την, τις υποδομές, να έχει ένα καλό σύστημα εκπαίδευσης Ε, αν είναι σημαντικό το να βρίσκεται κανείς κοντά στα κέντρα γνώσης ε, και καινοτομίας, ε, τότε είναι σημαντικό ο κόσμος να έχει, οι εργαζόμενοι να έχουν υψηλές δεξιότητες. Επίσης χρειάζεται ένα ισχυρό και σταθερό κοινωνικό κλίμα. Ξέρουμε ότι ο κοινωνικός διάλογος ε, μπορεί να αποτελεί πρόκληση. Φαίνεται στην Ευρώπη ότι ε, χρειάζεται πολύ χρόνο κλπ. Αλλά ε, στην Κίνα ή στη Λατινική Αμερική όπου θα πάω απόψε ονειρεύονται ένα τέτοιο σύστημα. Υπάρχουν λοιπόν δυσκολίες με ένα τέτοιο σύστημα. Για να έχει κανείς ένα λειτουργικό σύστημα κοινωνικού διαλόγου αποτελεί όμως σίγουρα ένα ατού της Ευρώπης. Υπάρχουν επίσης ε, πολιτικές που παίζουν ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι το ψυχιακό θεματολόγιο και το σχέδιο Juncker είναι πάρα πολύ σημαντικά εάν ε, προσανατολιστούν στο να κάνουν πιο ελκυστική την Ευρώπη. Και Εάν συνδέσουμε το θεματολόγιο αυτό με το θέμα των επενδύσεων, ε, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη. Οι επενδύσεις είναι ανεπαρκείς στην Ευρώπη. Αν εξετάσουμε τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, ε, παραμένει το ποσοστό αυτό ε, πιο κάτω από, από τα επίπεδα πριν την οικονομική κρίση και είναι σημαντικό το σχέδιο Juncker, υπάρχει όμως και έλλειψη θέσεων απασχόλησης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το σχέδιο Juncker να χρησιμοποιηθεί να συνδεθούν οι επενδύσει από το σχέδιο Juncker με την ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Επίσης, ε, νέε πηγέ ενέργειας, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια μπορεί να αποτελέσουν μακροπρόθεσμα ε, σημαντικό ατού ώστε να γίνει πιο ελκυστική η Ευρώπη. Αυτά λοιπόν τα θετικά που μπορούν να γίνουν. Υπάρχουν και πράγματα που πρέπει να αποφύγουν, τα οποία μπορεί να είναι αντιπαραγωγικά εάν θέλουμε να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις ή επιστροφή των θέσεων εργασίας. Θα πρέπει να αποφύγουμε ε, την, ε, υποβάθμιση, την κοινωνική υποβάθμιση με την ε, μείωση των αποδοχών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ναι, το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υποστηρίζει κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί να μπει κανείς στον πειρασμό για να προσελκύσει επενδύσεις. Μία μεγάλη κοινωνία με σταθερή μεσαία τάξη μπορεί να θεωρείται ασύμβατη με την ε, διατήρηση των ε, δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά θα πρέπει να το προσέξουμε. Επίσης, ε, άλλος πειρασμός στον οποίο θα μπορούσε να πέσει κανείς είναι ο φορολογικός ανταγωνισμός, δηλαδή να μειώσει τη φορολογία για να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Η, ε, τα, τα δεδομένα όμως δεν δείχνουν ότι αυτό είναι πετυχημένη μακροπρόθεσμη στρατηγική. Νομίζω ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερο να επενδύσει στην εκπαίδευσή της. Και τώρα που πραγματοποιούνται συζητήσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και άλλα μέρη του κόσμου όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Σημαντικό είναι να προστατεύσουμε τις επενδύσεις, αν όμως η προστασία αυτή είναι υπερβολική. Αυτό θα μειώσει τις ε, δυνατότητες να έχουμε μία σταθερή και δυναμική μεσαία τάξη, κάτι που αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας ε, της Ευρώπης. Ε, θα κλείσω εδώ, νομίζω ότι εξήγησα και το δεκαλεπτό μου. Ευχαριστώ. Thank you. Then I'll give ο κύριος Τόνι Καλντέιδα, διευθυντής του Καλντέιδα Limited. Είστε ένα παράδειγμα από τον πραγματικό κόσμο. Πείτε μας για το παράδειγμά σας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όντως από τον ε, κόσμο της αγοράς έρχομαι. Είμαστε μια μικρή εταιρεία στο Λίβερπουλ, στη Βρετανία. Um, Αυτό που θέλω να σας πω σήμερα είναι πώς γίνεται ήδη ο επαναπατρισμός των επιχειρήσεων. Στη σημερινή μου παρουσίαση θέλω να εξηγήσω λίγο τα, τις εταιρείες μου για να καταλάβετε το background της εταιρείας μου και γιατί γίνεται πανοπατισμός, γιατί φέραμε πίσω κάποιες θέσεις από την Κίνα, κάποιες δραστηριότητες μας από την Κίνα στη Βρετανία και ελπίζω να σας βοηθήσω να καταλάβετε κάποια πράγματα από την οπτική του επιχειρηματία συμβουλεύοντας και τις κυβερνήσεις ενδεχομένως με αυτά που κάνουμε. Να σας πω την ιστορία μας. Την εταιρεία την έφτιαξα το 1991. Γίναμε leader στην αγορά, ε, με μαξιλάρια κυρίως. Από μικρό μαγαζί έγινε leader όπως σας είπα. Το 2003 είχα ψηλή θέση στην Βρετανία. Το 2003 Πήγαμε σε κάποιες παγκόσμιες εκθέσεις και διαπιστώσαμε ότι η Κίνα θα έμπαινε εκείνη την εποχή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και η τιμή πώληση ε, στην Κίνα ήταν ε, χαμηλότερες από τις βρετανικές τιμές, από το βρετανικό κόστος. Η επιλογή μας ήταν απλή. Ή να πάμε στην Κίνα ή να κλείσουμε. Κάναμε τη στρατηγική επιλογή να ανοίξουμε μια κοινοπραξία στην Κίνα και να κλείσουμε ένα από τα δύο εργοστάσια μας στην Βρετανία. Το άλλο το κρατήσαμε. Η Βρετανική, το Βρετανικό εργοστάσιο επιβίωσε την, της παγκοσμιοποίησης κάνοντας μία στάνταρ κίνηση πολλών. Κάναμε, ανεβήκαμε, γίναμε upmarket εταιρεία με καλύτερη ποιότητα, γρήγορη ε, αντίδραση, κοντά στην αγορά, περισσότερες υπηρεσίες πριν και μετά την αγορά. Προσπαθήσαμε να δουλέψουμε με τοπικές επιχειρήσεις για να κερδίσουμε. Επίσης αποφασίσαμε να ανοίξουμε ένα γραφείο στη Νέα Υόρκη για το Caldera USA που πουλούσε προϊόντα και Βρετανίας και από το βρετανικό και από το κινέζικο εργοστάσιο. Η καμπή για μας ήταν το 2007-2008 όταν τελείωσε η πρώτη φάση της παγκοσμιοποίησης και ξεκίνησε η επόμενη φάση, το επόμενο στάδιο της παγκοσμιοποίησης. Τότε η παλήρια άλλαξε. Ξαφνικά οι τιμές στην Κίνα άρχισαν γρηγορότερα από ό,τι στη Δύση. Ως αποτέλεσμα τούτου η Ευρώπη έγινε πιο, γίνεται πιο ανταγωνιστική κάθε χρόνο. Κάτι που δεν το καταλαβαίνουν πολλοί Ευρωπαίοι πολιτικοί. Ότι δηλαδή η Ευρώπη γίνονται ανταγωνιστική για μεγάλα χρόνια, για πολλά χρόνια. Δείτε τις δύο διαφάνειες που έχω. Αύξηση του μισθού των ε, Κινέζων εργαζομένων, ενώ βλέπετε την ανατίμηση του Ιουάν τα τελευταία 10-15 χρόνια. Προσθέτοντας τους δύο αυτούς παράγοντες και διαπιστώνουμε ότι τα κινέζικα προϊόντα είναι ακριβότερα, από, πολύ ακριβότερα από ό,τι στο παρελθόν. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε ότι το κόστος εργασίας για μας ε, ανέβηκε τρελά στην Κίνα. Εμείς έχουμε το εργοστάσιό μας σε μια περιοχή κοντά στη Σαγκάη. Οι εργαζόμενοι μας είχαν αύξηση σε 10 χρόνια των μισθών τους κατά 400%. Όταν πήγαμε το 2003-2004 στην Κίνα, οι Κινέζοι εργαζόμενοι έπαιρναν το 10% των αντίστοιχων Βρετανών, ενώ τώρα είναι 30 με 40% ανάλογα με τις ισοτιμίες του νομίσματος. Στο γράφημα αριστερά βλέπετε την, κινέζικη οικονομία και το μισθό που λαμβάνει ένας Κινέζος. Δεν είναι σαφής η κλίμακα, αλλά η αύξηση είναι 240% στους κινέζικους μισθούς μεταξύ του 2000 και του 2012. Μετά ε, το 2012 έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Δεξιά είναι το κόστος παραγωγής αναμονάδα στην Ευρωζώνη που είναι επίπεδη. Άρα οι Κινέζοι εργαζόμενοι ε, αυξάνουν, το, το κόστος των Κινέζων εργαζομένων αυξάνει. Άλλος βασικός παράγοντας για τα κέρδη ήταν η ισοτιμία. Σε 7 χρόνια το ευρώ έπεσε κατά 30% σε σχέση με το ρεμίμπι που κάνει ακόμα πιο ανταγωνιστικά τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Και άλλοι παράγοντες έχουν γίνει, έχουν παίξει ρόλο, αλλά βλέπετε πόσο πιο ανταγωνιστική είναι τώρα η Ευρώπη από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Τι έκανε λοιπόν η Καλντέρα. Αντιδρούμε, αντιδρούμε στις εξελίξεις στην αγορά. Αποτέλεσμα είναι ότι φέραμε κάποιες δραστηριότητες μας στην Βρετανία, οπότε μειώνουμε τις δραστηριότητες μας στην Κίνα και επαναφέρουμε δουλειές στην Βρετανία. Προφανώς επειδή δουλεύουμε με πολλούς, πρέπει να δουλεύουμε με τον τρόπο που μας λένε. Κάποιοι ζητούν να τους παρέχουμε τα προϊόντα FOB Σανγκάι, άλλοι να τους παρέχουμε τα προϊόντα FOB ε, Liverpool, Ακολουθούμε την πορεία πάντως και η πορεία αυτή τη στιγμή είναι προς την Ευρώπη. Επιχειρήσεις όπως οι δική μου αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά ζητήματα και έβαλα κάποιες παρατηρήσεις εδώ που θεωρώ σημαντικές ούτως ώστε να ξέρουν οι βουλευτές. Σε πολλές χώρες όταν η παραγωγή έφυγε χάθηκε και η τεχνολογία η επαναφορά λοιπόν των δεξιοτήτων δεν είναι πάντα εύκολη. Ταυτόχρονα και πολλά προσόντα χάθηκαν. Γνώσεις δηλαδή. Αυτό που πολλοί δεν καταλαβαίνουν είναι η σημασία της αλυσίδας ε, τροφοδοσίας στην, ε, στον κλάδο. Όταν έφυγαν από τη Βρετανία οι κλωστιοφαντουργικές δραστηριότητε τις αρχές της δεκαετίας του 2000, έφυγαν και επιχειρήσεις που προμήθευαν προϊόντα ε, υφαντουργικού χαρακτήρα. Επίσης, υπάρχει ένα πρόβλημα χρηματοδότησης. Για πολλούς ε, τραπεζίτες το να ε, ε, ζητάς λεφτά από μια τράπεζα να, για να φτιάξει μαξιλάρια στο Λίβερπουλ μπορεί να μην θεωρείται για πολλούς πολύ καλές, ε, ε, μια πολύ καλή δραστηριότητα. Τι προσπαθώ να κάνω τώρα εγώ εδώ. Να βοηθήσω τους πολιτικούς σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις πλευρές, να καταλάβουν τι ζητούν οι μικρές επιχειρήσεις από τις κυβερνήσεις. Το πρώτο που προτείνω είναι να έχει υψηλούς στόχους η Ευρώπη να κάνει τη χώρα και την, την εταιρεία και την Ήπειρο το καλύτερο μέσο, το καλύτερο μέρος για να επιχειρείς, να ασκείς επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό απαιτεί οικονομική σταθερότητα και γιατί τα σταθερά οικονομικά Ιδίω δημόσια οικονομικά, επιτρέπει στους επενδυτέ να λαμβάνουν μακροπρόθεσμες αποφάσεις και τους διασφαλίζει ότι ο επαναπατρισμό θα είναι θετικός. Το είπε και ο κύριο Τόρε Το τμήμα του εντατικού κεφαλαίου είναι αυτό που πρέπει να ενισχυθεί. Επίσης, το επιχειρηματικό περιβάλλον πρέπει να είναι φιλικό προς τις επιχειρήσεις. Πρέπει να πείσουμε τις επιχειρήσεις ότι αξίζει να επιστρέψουν χρειαζόμαστε χαμηλή, απλή, ανταγωνιστική και δίκαιη φορολογική νομοθεσία. Όχι τις πολιτικές που να βουτήξουμε τον επιχειρηματή από το γείτονα, αλλά αντίστοιχα καθεστώτα. Νομίζω ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να συζητήσουν την κατάσταση. Καλό είναι το μοντέλο των ΙΠΑ. Είναι σημαντικό να... Το, το, του Ηνωμένου συγγνώμη. Είναι σημαντικό να λέμε φέρετε τις επιχειρήσεις σας πίσω στην πατρίδα σε Βρετανούς, αλλά μπορεί να είναι ε, κάποιες επιχειρήσεις που να θέλουν να εγκατασταθούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό μέσα στην νέα αγορά θα πρέπει να ενισχύεται. Οι πολιτικοί μπορεί να θέσουν τις προσδοκίες και να βοηθήσουν στην εκπαίδευση των καταναλωτών. Μα λένε διάφορα, μα πώ μπορεί να ανταγωνιστεί στην Κίνα που είναι φθηνότερη. Εγώ πιστεύω ότι σε πολλού τομεί μπορούμε να την ανταγωνιστούμε και αν μια ευρωπαϊκή επιχείρηση μπορεί να, να γίνει ανταγωνιστική με την Κίνα, Τώρα, το σημείο της καμπής, αυτό που είναι το σημείο που αποφασίζει ο επιχειρηματίας να επαναπατρίσει την επιχείρησή του, μπορούν οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις να πείσουν τους ε, επιχειρηματίες να τις γυρίσουν στην πατρίδα τους και να βοηθήσουν στις Αλλά από τη στιγμή που φέρνεις επιχειρήσεις πρέπει να φέρεις όλη την αλυσίδα τροφοδοσίας. Έτσι, δεν δημιουργούνται μόνο θέσεις εργασία από την ίδια την επιχείρηση, αλλά και στην αλυσίδα. Εγώ, για παράδειγμα, η δική μου επιχείρηση έχει φέρει πολλές νέες θέσεις εργασίας άσχετες άμεσα με την επιχείρηση, σχεδιαστές, ε, δεν, είναι δηλαδή, δεν μόνο οι κατασκευαστικές ε, θέσει εργασία, αλλά και οι συναφείς. Κάτι πολύ σημαντικό. Επίσης, οι επενδύση είναι βασικός παράγοντας. Η εκπαίδευση θα βοηθήσει να επανέλθουν κάποια από τα προσόντα που χάθηκαν. Η παροχή κινήτων σημαίνει να καταλάβουμε, να βοηθήσουμε τις να καταλάβουν για το πώς θα ξαναφέρουν πίσω τις επιχειρήσεις. Γιατί πάρα πολλές φορές ένας Ευρωπαίος επιχειρηματίας προτιμά να το κάνει σπίτι του, στην πατρίδα του αυτή τη δουλειά από το εξωτερικό. Αυτό που επίσης πρέπει να καταλάβουν τα μέλη σήμερα είναι ότι η ευκαιρία είναι εν δυνάμει τεράστια αν το υφιστάμενο μοντέλο μείωσης υποτίμησης, ε, ανατίμησης του, του και αύξησης των εισοδημάτων και των αμοιβών των ε, Κινέζων εργαζομένων σημαίνει ότι θα γίνει τώρα και λιγότερο ανταγωνιστική η Κίνα. Για την ε, αμερικανική θηγατρική μας είναι σημαντικό να προχωρήσει και το TTIP. Έχουμε αντικαταστήσει προϊόντα αμερικανικά με ευρωπαϊκά υφάσματα που γίνονται στην, ε, στη ΣΥΠΑ. Αν αυτό μπορούμε να το κάνουμε με λιγότερη γραφειοκρατία θα δημιουργηθούν επίσης και νέε θέσει εργασία στην ε, Βρετανία και θα δημιουργηθεί και την Ευρώπη και θα δημιουργηθεί ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον. Ένα τελευταίο τελικό θέμα. Εγώ πιστεύω ότι σας είπα ότι γίνεται, υπάρχει αυτή τη στιγμή επαναπατρισμός, γίνεται. Το ερώτημα πάντως που θέτω στους βουλευτές σήμερα είναι είστε έτοιμοι για τον επαναπατρισμό. Κάποιε χώρες δεν είναι νομίζω. Πρέπει λοιπόν να έχετε επίγνωση ότι αυτό το γεγονό συμβαίνει και όποιος το καταλάβει γρήγορα θα κερδίσει περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καλτέρα και τώρα θα πάρει το λόγο ο κύριος Μανουέλ Γκαρσία Σαλγάδο που είναι ε, ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Νομοσπονδίας Εργατών της Χαλιβουργίας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Γεια σας. Χαίρομαι που είμαι εδώ στην Επιτροπή σας. Τα παραδείγματα που εγώ έχω πηγαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Είχαμε, θα σας κάνω μια παρουσίαση της αλλαγής του εργασιακού χάρτη στην Ισπανία, του, της εργασιακής νομοθεσίας στην Ισπανία του Φεβρουαρίου που έγινε μετά από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και που κατόπιν η ίδια η Επιτροπή την ενέκρινε η κυβέρνηση που την εφάρμοσε πέταξε το προεκλογικό της πρόγραμμα στα σκουπίδια και έβαλε, έκανε αυτό που της είπε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα δούμε τώρα τις συνέπειες πρώτα άμεσα και μετά ευρύτερα. Πρώτη συνέπεια, σημαντική μείωση της ε, συμμετοχής στο ΊΚΑ στην κοινωνική ασφάλιση. Από το 2011 μειώθηκαν 400, οι θέσει εργασία κατά 423.000 παρά τη μεταρρύθμιση που υποτίθεται ότι έγινε για να δημιουργηθούν θέσει εργασία. Μία στι τέσσερι θέσει εργασία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ισπανία έχουν προσωρινό χαρακτήρα, υποχρεωτικά προσωρινό γιατί δεν υπάρχει άλλη προσδοκία δουλειά. Δηλαδή, εδώ μιλούμε για νέου. Ένα στους τέσσερις νέους δουλεύουν ε, ώρα με ώρα. Με ώρες, όχι με ημέρες, όχι με μισθό. 23% είναι ακόμα και σήμερα με προσωρινά ή επισφαλή, ε, με προσωρινές επισφαλείς συμβάσεις εργασίας. ανεβαίνει σημαντικά η, απασχόληση, η μερική απασχόληση. Το ποσοστό των εργαζομένων με μερική απασχόληση είναι 16,3%. Αλλά πάνω από 61% από αυτούς το κάνουν χωρίς να το θέλουν. Απλώς δεν βρίσκουν άλλη δουλειά. Έγινε λοιπόν ένα διαρθρωτικό στοιχείο της ε, ισπανικής αγοράς εργασίας. Όπως σας είπα, ένας εργαζόμενος στους τέσσερις δουλεύουν με προσωρινές συμβάσεις. Το 23,6% πιο συγκεκριμένα. Η ανεργία στην Ισπανία αυτή τη στιγμή πλήττει έναν στους τέσσερις εργαζόμενους. Και αυτό σύμφωνα με τις έρευνες ενεργού πληθυσμού, δηλαδή αυτών που είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν αλλά δεν μπορούν να το κάνουν. Αυτό ο πίνακας δημοσιεύτηκε φέτος τον Ιούλιο. ...22,37% είναι η ενεργεία σήμερα. Αυτό οδήγησε σε φτώχεια των εργαζομένων, ατόμων που μερικέ φορέ έχουν και δουλειά και παρόλο που έχουν δουλειά δεν μπορούν να καλύψουν τη βασική, τις βασικές τους ανάγκες. Άρα υπήρξε σημαντική αύξηση της φτώχειας και μιλούμε για 20% φτώχεια. η ανεργία των νέων ε, παραμένει ψηλή, ψηλότερη και από πριν τη μεταρρύθμιση. Τον Ιούλιο φέτος ήταν σχεδόν το 50%. 49,2 ειδικότερα. Των νέων κάτω των 25 που βρίσκονται σε ανεργία. Χωρίς να λάβουμε υπόψη τη μεγάλη μετανάστευση που είχαμε προς άλλες χώρες της Ευρώπης και αλλού. Και το σημαντικό ποσοστό μεταναστών στη χώρα μου που χρειάστηκε να φύγουν και να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. το ποσοστό των ε, μακροχρόνιων ενεργών άνω του 1 και των 2 έτος και των 2 ετών αυξήθηκε σημαντικά. Σήμερα υπάρχουν εργαζόμενοι, πολλοί εργαζόμενοι που δεν έχουν πλέον καμία, κανένα επίδομα. Ενώ ταυτόχρονα διπλασιάστηκε ο αριθμό των ε, μακροχρόνιων ενέργων. Άρα το επόμενο βήμα είναι ο κοινωνικός Αποκλεισμό ατόμων που δεν έχουν καμία προσδοκία να επανέλθουν στην αγορά εργασία. Αυτό είναι το γράφημα που αποδεικνύει αυτή την εξέταση. Το ποσοστό αυτών που δεν λαμβάνουν επιδόματα είναι μεγαλύτερο, ενώ το ποσοστό κοινωνικής κάλυψης λόγω ανεργίας ε, ανέβηκε και μετά ξαναμειώνεται. Οι συμβάσεις εργασίας ε, κρατούν δύο μήνες λιγότερο, ακόμη και σε τομείς που δεν είχαν ε, τον ευάλωτο χαρακτήρα των θέσεων εργασίας, δηλαδή η βιομηχανία κυρίως που είναι αυτή που δημιουργεί το μεγαλύτερο ρυθμό σταθερών ε, θέσεων εργασίας με δικαιώματα σε μεγαλύτερη συμμετοχή στα ταμεία και διαθροτικές επιπτώσεις έγινε και αυτός ο κλάδος ευάλωτων εργαζομένων. Εδώ βλέπετε αυτό το πράγμα. Οι προσωρινές συμβάσεις ε, είναι 91% για, την, ε, για τον κλάδο της μηχανίας και 85% για τον κλάδο της, ε, των υπηρεσιών. Ανέβηκε δηλαδή σε σχέση με παλαιότερα. Ένας, μία, μία στις τέσσερις συμβάσεις των κλάδο έχει διάρκεια μικρότερη από 7 μέρες. Από 7 έγινε 24%. Επίσης, ε, δημιουργήθηκε η, η έννοια της εποχιακής εργασίας και σε μια μέρα τέλη Αυγούστου πέρσι απολύθηκαν 333.000 άτομα. Ποτέ άλλοτε δεν έγινε κάτι τέτοιο στην Ισπανία. Γιατί, διότι πάρα πολλές ε, θέσεις είναι προσωρινές, ε, ευάλωτες, δεν υπάρχει ένα οικονομικό μοντέλο που δημιουργεί σταθερή δουλειά και το γεγονός ότι μπορείς να απολύεις τον κόσμο από το ίντερνετ, μέσω ίντερνετ δηλαδή, μέσω το Σαββατοκύριακο, για να μην πληρώνεις το Σαββατοκύριακο. Κάτι που δημιουργεί ένα χάος στην αγορά εργασία, περισσότερο από το υφιστάμενο. Εναλλακτικέ και προτάσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι για να αλλάξει η κατάσταση αυτή και να γίνει η Ευρώπη ένα κοινωνικό μοντέλο πραγματικό, ισορροπημένο, με δικαιώματα, που θα είναι ανταγωνιστική δεν μπορεί να γίνει μέσω φυσιολογικών μειώσεων. Αυτό που σας να κάνει η μεταρρύθμιση στην Ισπανία. Προφανώς πάντα θα υπάρχουν χώρες και περιοχές στον κόσμο που θα είναι φτηνότερες από την Ευρώπη. Το Παγκλαντές, το Πακιστάν, μια άλλη χώρα εμείς θεωρούμε ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο πρέπει να είναι άλλο. Να βοηθά στην ενίσχυση μιας ενεργής βιομηχανικής πολιτικής και σε επίπεδο κράτους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι η πρόταση που έκανε στο Κοινοβούλιο η Ένωση Ευρωπαϊκών Συνδικάτων την προσέγγιση αυτή πρέπει να συμπεριλαμβάνονται παράμετροι που στηρίζονται στην περιβαλλοντική βιομηχανία, την καθαρή ενέργεια, την έρευνα και την επένδυση στην έρευνα και, και ανάπτυξη, την ε, δημιουργία υποδομών, τον κοινωνικό διάλογο, τη συλλογική διαπραγμάτευση και την εναρμόνιση, την προοδευτική εναρμόνιση των εργατικών, της εργατικής νομοθεσίας τεράστιος πολιτικός και νομισματικός χώρος. Ας προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση σαν να είμαστε εργαζόμενοι στον ίδιο πολιτικό χώρο. Επίσης δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ότι χωρίς επένδυση στην παιδεία και την εκπαίδευση, χωρίς δηλαδή ε, επένδυση στην καινοτομία ως προστιθέμενη αξία, δεν θα αναδείξουμε την, ε, πρώτο, την υπεροχή της Ευρώπης στον υπόλοιπο κόσμο. Αν η Ευρώπη αλλάξει το μοντέλο της, προχωρήσει προς την μείωση των δικαιωμάτων και ε, δεν κάνει ένα διάλογο με τα διάφορα μέρη, θα χάσει το βασικό λόγο της. Στις ανταγωνιστικές κοινότητες και εκεί όπου υπάρχει μια μεγαλύτερη συμμετοχή και συνεισφορά των εργαζομένων στις ε, παραγωγικές διαδικασίες, στην βελτίωση και στην καλύτερη γνώση της επιχείρησης του καθενός στο κομμάτι που αντιστοιχεί στον καθένα διότι αυτός είναι ο πρώτος ο οποίος θέλει να φτάσει στην οικογένειά του μια μέρα πριν Η υποτίμηση της ε, αξίας εργασίας δημιουργεί φτωχούς, δεν δίνει θέση εργασίας και δεν διευκολύνει την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας προς μια παραγωγική οικονομία που θα βασίζεται στην επένθυση και την οικονομική και κοινωνική συνεργασία. Αυτά είναι γενικά οι Δηλαδή τα βήματα που κάνουμε. Το σχέδιο Χιούνκερ είναι καλό αρχιεραρχικές ε, πλάνο. Το ευρωπαϊκό μοντέλο πρέπει να βασίζεται στις κοινωνικές συνθήκες ισορροπίας και προστασίας των ατόμων για να μπορέσουν να διευκολύνουν τον άνθρωπο να κάνει μια αξιοπρεπή ζωή. Δεν μπορεί να έχουμε ανέργους άτομα που αντιστοιχούν στο τέταρτο του πληθυσμού, άνθρωποι που πρέπει να που γνωρίζουν την κατάσταση θα πρέπει να ξέρουν ότι αυτό σημαίνει αποκεφαλοποίηση του, της οικονομίας. Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για τις εισαγωγικές σας παρεμβάσεις. Δεν ήταν πολύ αισιόδοξα αυτά που μας είπατε, αλλά Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε ρεαλιστικά και να δούμε που θα καταλήξουμε. Κάποιοι από εσά ήδη ζήτησαν το λόγο. Δίνω πρώτα το λόγο στην... στον Έτου Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ στους τρεις ε, ομιλητές είναι τρεις ε, μαρτυρίες, ε, τρεις εισηγήσεις που μας δίνουν, ε, δείχνουν βασικά ότι δεν θα έπρεπε να είναι η Ευρώπη. Και είμαι περήφανος που άκουσα τον πρώτο μας καλεσμένο που μας μιλά για το κοινωνικό διάλογο έχει στιγματιστεί ο κόσμος της εργασίας και έχει πληγωθεί επίσης. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για να έρθουν οι εταιρείε να εγκατασταθούν στην Ευρώπη. Και σας ευχαριστώ. Ήσασταν πάρα πολύ καλοί ε, ε, πολιτές για την Ευρώπη, για το ευρωπαϊκό κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο. Είναι ένα επιχείρημα ε, προσέλκυσης, ε, το να υπάρχει σταθερότητα οικονομική ή κοινωνική ε, θα έπρεπε να ελκύει όντως τις επιχειρήσεις. Όμως ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, όμως εδώ δυστυχώς δεν είναι λεπτομέρεια. Έχουμε πέσει στην παγίδα που πολλοί μας έχουν στήσει ότι αυτή η περίφημη ανάκαμψη δεν θα έρθει παρά μόνο μέσω της ε, καταπολέμησης της, του, αγώνα κατά του κόστους της εργασίας, ε, όπως στην Ισπανία που έχουν καταστραφεί τα δικαιώματα των Ισπανών και ορισμένοι θριαμβολογούν και λένε και ξαναλένε ότι η Ισπανία πάει καλύτερα. Ποια η Ισπανία πάει καλύτερα, των πλούσιων, η Ισπανία όμως των εργαζομένων και ο συνάδελφος μας το απέδειξε έχει ε, διαλυθεί. 50% ανεργία στους νέους. Αυτό θα πει ότι πάει ωραία η Ισπανία, είναι κανείς περήφανος γι' αυτό. Όλες οι συμβάσεις εργασίας είναι κάτω των δύο μηνών, αν αυτή είναι η προπτική της Ευρώπης, προφανώς θα είναι χωρίς εμάς. Και εγώ υποστηρίζω την καταδίκη που προέφερε ο συνάδελφός μας ε, από το συνδικάτο και θέλω να καλέσω την Ευρώπη να τα, πάει, να τα κάνει διαφορετικά τα πράγματα. Το είπε και πρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας και ο κ. Καλδέρα ότι έχουμε ατού έχουμε πλανεκτήματα, είμαστε, είμαστε πιο ανταγωνιστικοί γιατί έχουμε διαρκή ας πούμε κατάρτιση και αυτό υπόθηκε και υπογραμμίστηκε. Είναι αυτό το κεφάλαιό μας, ε, οι δεξιότητες, οι ικανότητες, αντίθετα από το ισπανικό πρότυπο, όταν κανείς ε, ενθαρρύνει και γενικεύει την επισφάλεια, ολόκληρη η ε, ανταγωνιστικότητα της χώρας θα γίνει, θα, θα γίνει μάλλον αισθητό αυτό πραγματικά σε ολόκληρη τη χώρα. Γιατί δεν θα βρεις κανέναν τεχνικό ε, προσόντα όταν θα το χρειαστεί, γιατί θα έχουμε καταστρέψει το ανθρώπινο κεφάλαιό μας. Εγώ θα έλεγα ότι η κρίση είναι κρίση επενδύσεων και πρόσβαση στις πιστώσεις. Και εδώ η Ευρώπη πρέπει να αποκομίσει τα διδάγματα των τελευταίων ετών κρίση και να καταλάβει ότι πάει ανάποδα. Δεν μπορεί να συνεχίσει πια έτσι και το υπογράμμισε και ο εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού ε, εργασία ότι όλε οι πολιτικέ αυτές γίνονται υποτίθεται για να εξασφαλίσουν τι επενδύσει και να το υπερασφαλίσουν τι επενδύσει στην ε, ΣΥΠΑ και σε αυτόν τον κόσμο ζούμε. Δηλαδή όλε οι πολιτικέ που κάνουμε και το σχέδιο Juncker μαζί, τι θέλουν να καθησυχάσουν τον επενδυτή. Ναι, ελάτε να επενδύσετε εδώ, δεν θα, δεν θα κινδυνεύσετε τίποτα, γιατί, γιατί οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που θα ζήσουν στην επισφάλεια, αυτοί που θα ζουν με αβεβαιότητα συνέχεια, θα τους καταργήσουμε τα κοινωνικά τους δικαιώματα και ούτω καθεξής. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται πλέον. Ευχαριστώ και τον κύριο Καλτέρα για τα όσα μας είπε ότι η Ευρώπη ναι μπορεί να είναι πιο ανταγωνιστική με την προϋπόθεση να διατηρήσει τις αξίες της και το είπατε δηλαδή επενδύσεις στις υποδομές, κατάρτιση, παιδεία Λυπούμε μόνο ότι δεν έγινε, που δεν έγινε αρκετός λόγος για την περιβαλλοντική Ευρώπη, για το κλίμα που ήδη είναι όλο ένα και περισσότερο επίσης ένας ε, παράγοντας ανταγωνιστικότητας και πιστεύω ότι οι θέσεις που υπερασπιζόμαστε ώστε η Ευρώπη να διατηρήσει αυτά τα πλεονεκτήματα όσον αφορά το περιβάλλον, ανανεώσιμε πηγές ενέργεια, είναι επίση ένας τομέας για να βοηθήσουμε να μετεγκατασταθούν, να επανέλθουν, επαναπατριστούν πολλές εταιρείε. Ευχαριστώ και πάλι τους τρεις ομιλητές μας. I give the floor to Madam McIntyre. Η κυρία Μάκιντάιρ τώρα. Thank you very much, uh, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Συναρπαστικές και οι τρει εισηγήσεις. Είμαι ευγνώμων στον κύριο Τόρε που μας έδωσε κάποια στατιστικά στοιχεία και που τόνισε τις πιθανές τάσεις, ακόμα κι αν δεν έχουμε ακόμα επιστημονικές αποδείξεις, τονίσατε τις τάσεις ότι η περισσότερη παραγωγή γίνεται στην Ευρώπη αντί εκτός, αλλά ότι, και ότι, χρειάζονται περισσότερο, ότι έρχονται περισσότερες επενδύσεις εντός της Ευρώπης από ότι εκτός της Ευρώπης. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Επίσης, ε, πολύ μου άρεσε που άκουσα από τον Τόνι Καλτέρα την επιτυχία της εταιρείας του, και τον τρόπο με τον οποίο μπόρεσε να επαναπατρίσει θέσεις στην Ευρώπη, σε αυτή την περίπτωση, πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πιστεύω πως το μανιφέστο του για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στο να συνεχιστούν όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέρον. Εσείς κύριε Σαλγκάντο όμως με απογοητεύσατε. Με στεναχωρήσατε. Στεναχωριέμαι πολύ για την Ισπανία. Γιατί εκεί που ζω εγώ, βλέπουμε αύξηση των θέσεων απασχόλησης και βλέπουμε επίσης ότι η ανάπτυξη είναι 2,8% στην απασχόληση. Ε, περισσότερος κόσμος αρχίζει να δουλεύει και πραγματικά με λυπεί που η δική σας εμπειρία στην Ισπανία είναι έτσι. Γιατί πρέπει να σας πω ότι δεν είναι υποχρεωτικό να πάνε έτσι τα πράγματα. Αν κατανοούμε την σημασία της βοήθειας προς τους επιχειρηματίες, ε, να, μην τους ε, καθυστερούμε, να μην τους ε, μπλοκάρουμε με γραφειοκρατία. Μπορούμε να βοηθήσουμε λοιπόν τις εταιρείε που θέλουν να επαναπατρίσουν θέσεις στην Ευρώπη. Εγώ είμαι οπαδός του Αντιπροέδρου Τίμερμαν της Κομισιόν, γιατί αυτός είναι σοσιαλιστός. Εγώ είμαι συντηρητική, αλλά είναι σοσιαλιστής και εγώ συμφωνώ πολύ με την προσέγγιση του και την ιδέα του για καλύτερη νομοθεσία. Γιατί έτσι μπορούμε να διευκολύνουμε τους επιχειρηματίες μας να κάνουν περισσότερο χρόνο τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Θα θυμάστε συνάδελφοι τα παραδείγματα που είχαμε του φούρναρη που πρέπει να μπορεί να κάνει περισσότερη ώρα στο φούρνο φτιάχνοντας ψωμί παρά να συμπληρώνοντας ε, ε, έντυπα και δελτία. Πώς λοιπόν πιστεύετε ότι αυτή η υπόθεση της καλύτερης νομοθεσίας μπορεί να βοηθήσει με την ε, υπόθεση της ε, εξασφάλισης και επίση για την καινοτομία. Ξέρω πολύ καλά ότι πρέπει να προσέξουμε ως νομοθέτες να μην πνίγουμε την καινοτομία. Δηλαδή, μπορεί να, να διευκρινίσουμε το τι θέλουμε να πετύχουμε, αλλά όχι το πώς απαραίτητος ας πούμε, αν είσαι πολύ, πολύ συγκεκριμένο στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνουν τα πράγματα, δεν επιτρέπει ένα χώρο για την καινοτομία και την νέα σκέψη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε θετικά το πρόγραμμα Ορίζοντας 2000 και έχουμε και 80 εκατομμύρια ε, ευρώ σε πέντε χρόνια. Και ένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του προγράμματος είναι ότι δεν είναι μόνο έρευνα, γενική και αόριστη, αλλά ότι πρέπει να ε, είναι και πρακτική εργασία σχεδιασμού και καινοτομία ώστε να φτάνει και στις μικρές επιχειρήσεις και να μπορούν αυτές να το χρησιμοποιήσουν. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, με την καινοτομία, θα βοηθηθούν να είναι πιο ανταγωνιστικοί. Και αυτό θα τις θέσει και στην πρωτοπορία και καθιστά πιο πιθανό το να επαναπατριστούν θέσεις απασχόλησης που παλιότερα ε, είχαν ε, φύγει. Εγώ πιστεύω πως το μέλλον είναι λαμπρό και θα ήθελα να ακούσω από τους τρεις μας ομιλητές ε, τη γνώμη τους για τα όσα είπα. Ναι, θα ξαναπάρουν τον λόγο. Στον κατάλογο μας τώρα είναι η κυρία και η Μαρία Ρένα, ο κ. Μπαλάς και η Μαρτίνα Λάγιουβα. Η κυρία Στάινμπροκ πρώτα. Καταρχάς να ευχαριστήσω και τους τρεις ομιλητές που βρήκαν το χρόνο να συζητήσουν εδώ μαζί μας το θέμα αυτό. Πρωτού πολιτικός, κινούμουν σε έναν κόσμο επιχειρήσεων, όπου έβλεπα τις επιχειρήσεις να εγκαταλείπουν την Ευρώπη για να μετακατασταθούν στην Ασία και πολύ συχνά από την Ασία μετά στην Αφρική. Για να είναι φθηνή η παραγωγή. Προσανατολίζονταν δηλαδή στο χαμηλό ε, κόστος μισθοδοσίας. Η Νόκια είναι ένα παράδειγμα. Η Ευρώπη καλά θα έκανε να αναλάβει σε περιφερειακό επίπεδο την ευθύνη. Υπάρχουν κάποια καλά παραδείγματα. Νομίζω ότι κάποιος από τους ομιλητές ε, το είπε ότι φθηνή παραγωγή πάντα θα υπάρχει αλλού στην, στον κόσμο, αλλά χρειαζόμαστε ανταγωνιστικότητα και όσον αφορά τις δεξιότητες και όσον αφορά την ε, τεχνολογία και την εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε δημόσιες επενδύσεις οι οποίες πληρώνονται από τον φορολογούμενο, δηλαδή και από τις επιχειρήσεις. το μέλλον. Όλα αυτά θα χρηματοδοτούνται από την φορολογία. Έτσι λοιπόν έχουμε τη ζυγαριά. Όποιος ε, δεν θέλει ε, όποιος δεν θέλει μετακατάσταση των επιχειρήσεων ε, θα πρέπει ε, να πληρώνει για να δημιουργηθεί ένα θετικό περιβάλλον. δεν επιτρέπεται να βλέπουμε μόνο τη μία πλευρά, θα πρέπει πάντα να έχουμε τη συνολική εικόνα. Όταν κοιτώ την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ε, σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των ε, μισθών, νομίζω ότι έχουμε ανέβει. Κύριε Καλτέρας, χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ. Τα αυτοκίνητα δεν αγοράζουν αυτοκίνητα, οι εργαζόμενοι τα αγοράζουν. Ε, θα πρέπει λοιπόν και σε αυτό το σημείο να φροντίσουμε να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία. Να επιτρέπουμε δηλαδή στους καταναλωτές να βγάζουν αρκετά λεφτά για να ε, μπορούν να αγοράζουν προϊόντα. Ίσως θα μπορούσαν και οι τρεις ομιλητές να αναφερθούν στο θέμα αυτό. Κύριε Καλδέρα, είσαστε παράδειγμα μιας επιχείρησης που επέστρεψε. Θα ήθελα να ρωτήσω, επανήλθαν εξίσου πολλές θέσεις εργασίας όσες μετεκαταστάθηκαν τότε εκτός Ευρώπης. και γνωρίζετε άλλα τέτοια παραδείγματα. Και υπάρχουν και επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, κάτι που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό μας. το παράδειγμα της Ισπανίας. Αναφερθήκαμε στην βιομηχανία μετάλλων, υπάρχει η βιομηχανία αυτοκινήτων, υπάρχει, ε, υπάρχουν άλλοι τομείς. Ε, θα ήθελα συγκεκριμένα παραδείγματα. Το, ο Διεθνής Οργανισμός ε, Εργασίας επίσης έχει κάποια στοιχεία, αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε σήμερα εδώ ένα ζωντανό παράδειγμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μαρία Ρένα. Ευχαριστώ. Τελικά θα, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει αυτή την ε, ε, ακρόαση μαζί με την Επιτροπή Ίντα, γιατί περισσότεροι μιλήσατε ταυτόχρονα για την πραγματικότητα, για την ε, επανεγκατάσταση στην Ευρώπη, αλλά και για τον αντίκτυπο επίσης της παγκοσμιοποίησης, γιατί είμαστε σε πολύ κατακαιρματισμένες αλλά και παγκοσμιοποιημένες ταυτόχρονα οικονομίες, οπότε η ελεπίδραση είναι σημαντική. Εγώ είμαι και στις δύο επιτροπές, οπότε μπορώ να μιλήσω και για την ΙΝΤΑ και για την ε, Επιτροπή ε, Απασχόλησης και συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε η Γιώτα. Κύριε μας εκφράσατε τη δυσκολία που έχετε να συμμορφώσετε ας πούμε την Κίνα με τον ε, ΠΟΕ αλλά ταυτόχρονα ε, μας είπατε πόσο θέλετε να, πόσο, πόσο είστε μάλλον υπέρ της υπερατλαντικής συμφωνίας ενώ άλλοι λένε εγώ μια χαρά θέλω την Κίνα μέσα στον ΠΟΕ. Αντίθετα, το που θα μου δημιουργήσει πρόβλημα θέμη του ανταγωνισμού. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε ακούσει κάποιον τελείως ε, ε με τελείως αντίθετη άποψη από τη δική σας. Τι κάνουμε εμείς τώρα με όλα αυτά. Και αυτό την ερώτηση θέλω να θέσω και στο Παγκόσμιο Οργανισμό Απασχόληση. Δουλεύουμε μέσα στο πλαίσιο αυτή τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών και θέλουμε οπωσδήποτε να μπει στην ημερήσια διάταξη και το θέμα τη βιώσιμη και σταθερή ανάπτυξη. Δηλαδή, οι κανόνε του Διεθνού Γραφείου Εργασία, του Διεθνού Οργανισμού Εργασία, όλα αυτά τα πρότυπα που είναι πρότυπα στην ουσία ευημερίες ε, για το περιβάλλον και για την κοινωνία όλα αυτά να μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτές τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, ούτως ώστε ο αθέμητος ανταγωνισμός που εσείς κύριε Καλτέρα καταγγέλλετε, αλλά θα μπορούσε κάποιος, κάποια άλλη εταιρεία να την καταγγείλει με τη ΣΥΠΑ, να μην ισχύει πλέον. Να, αυτές οι συμφωνίες, οι εμπορικές, να μην είναι πια συμφωνίες αθέμητου ανταγωνισμού. Γιατί σήμερα αυτό που έχουμε είναι εμπορικές συμφωνίες που είναι συμφωνίες αθέμητου ανταγωνισμού και που υπό την ε, κάλυψη μιας υποτιθέμενης πιο εύκολης νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις είναι στην ουσία μια απορρίθμιση και δεν συμφωνώ απόλυτα, εμένα μου αρέσουν οι κανόνες που προστατεύουν τον κόσμο. Καλύτερη νομοθεσία δεν σημαίνει μη νομοθεσία, απουσία νομοθεσίας και πολλές φορές ε, μάλιστα έρχομαι σε αντίθεση με τον κύριο Τίμερμανς, ακόμα και αν είναι σοσιαλιστός, όταν ακριβώς συχαίωμε το better regulation με το no regulation, την καλύτερη νομοθεσία με την καθόλου νομοθεσία. Ας πούμε, μιλάμε για την... Ε, ε, συμφωνία Ελευθέρων συναλλαγών, συναλλαγών για τις υπηρεσίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει απορρίθμιση των υπηρεσιών. Όλο ένα πιο ψηφιακά γίνονται όλα αυτά, αλλά δεν υπάρχει κανένας κανόνας. Κοιτάξτε τι γίνεται με το Uber, με στον τομέα του ταξί η απουσία κανόνων και το γεγονό ότι μια Αμερικανική εταιρεία κερδίζει λεφτά με βάση την καταστροφή του ευρωπαϊκού προτύπου δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Χρειάζονται κανόνε όταν γίνεται λοιπόν διεθνέ εμπόριο. Και θέτω το ερώτημα στο Διεθνή Οργανισμό Εργασία. Εσείς είστε υπέρ τη δέσμευση, τη δεσμευτικότητα αυτών των κανόνων γιατί έτσι μόνο μπορούμε να προστατεύσουμε τα δικά μας πρότυπα. Ευχαριστώ, Ματίνα Διαμπάλοβα. Πρέπει να σας πω ότι εγώ προσωπικά και η Άλντε Γέννη είμαστε υπέρ όντως της επιστροφής. Υπάρχει μια νέα ευκαιρία του επαναπατρισμού, υπάρχει μια νέα ευκαιρία για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους νέους. Απλά θα ήθελα να πω κάτι που είπε ο κύριος Καλδέρα ότι έρχεται από τον πραγματικό κόσμο και εγώ στον πραγματικό κόσμο ήμουν μέχρι πριν από ένα χρόνο και κάτι και προσέφερα υπηρεσίε στις μεταπητικές εταιρείε που χρειάζονταν νέες διεθνείς στρατηγικές ήταν ενδιαφέρον γιατί τα τελευταία 20 χρόνια είδα την Ευρώπη να αλλάζει. Καταρχήν οι εταιρείε από τις αρχές του 1990 μετακινούνταν από την Δυτική Ευρώπη στην Ανατολική λόγω των ε, πλεονεκτημάτων ε, όσον αφορά το κόστος ε, της εργασίας, το κόστος, το κόστος των κτηρίων. Μετά μετακινήθηκαν σε άλλες αγορές εκτός Ευρώπης, αλλά για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά. Στην αρχή ήταν συγκριτική διαφορά του κόστους, μετά ήταν η πρόσβαση στις νέες αγορές, γιατί ήταν στρατηγικό το να είναι κανείς αλλού και να έχει πρόσβαση σε νέε αγορές και λόγω της ευέλικτη αγορά εργασία, γιατί σε κάποια κάτι μέλη στην Ευρώπη δεν έβρισκαν την ευελιξία της αγοράς που χρειάζονταν. Οπότε πήγαιναν κάπου αλλού και ορισμένες φορές ε, ε, μετακινούνταν λόγω εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού. Δεν έβρισκαν το κατάλληλο εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη. Υπάρχουν διαφορετικοί ε, λόγοι λοιπόν και κάθε εταιρεία έχει διεθνή, διαφορετική διεθνή στρατηγική. Πρέπει άρα να εξετάσουμε το θέμα από διάφορες μεριές. Όμω να σας πω κύριε Καλτέρα, μην σταματάτε να μιλάτε περισσότερο στους πολιτικούς για τις ανάγκες σας, για τις ανάγκες των μικρομεσαίων ε, των μεταπητικών μηχανιών γιατί το χρειαζόμαστε, χρειάζεται να ενημερωνόμαστε συνέχεια για το τι συμβαίνει και για το τι χρειάζονται οι επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πιο, σημα... το πιο σημαντικό για μένα που θα ήθελα να ξέρω τη γνώμη και των τριών ομιλητών Μιλήσαμε για διαφορετικό κόστος, για νέες αγορές, για ευέλικτη αγορά εργασίας, για ειδικευμένο προσωπικό εργατικό δυναμικό. Κατά τη γνώμη σας αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να προσφέρει περισσότερα από ό,τι άλλες αγορές. Και τι ακριβώς, σε ποιο τομέα, είναι το εκπαιδευμένο προσωπικό, είναι ο ωραίος καιρός, δεν ξέρω. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας το ατού της Ευρώπης, κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να προωθήσουμε για να πουλήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερη παρατήρηση, και εδώ συγκεκριμένα στον κύριο Καλδέρα. ποιε είναι οι καλέ σα πρακτικέ για τους νέους. Ε, υπάρχει κάτι, κάποια ειδική στρατηγική με μαθήτιες, καταρτήσεις και κατά πόσο αυτό καθησυχάζει του επενδυτές. Και άλλη μια ερώτηση για τους τρει σα. Τι είδους μέτρα θα προτείνατε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να ε, οθήσουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη όταν ε, λειτουργούν εδώ στην Ευρώπη. Τι μέτρα έχετε στο μυαλό σας και τελευταία παρατήρηση που θέλω να τονίσω και το ανέφερε ο πρώτος ομιλητής αυτό και με ευγνώμων που το αναφέρατε είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει η Ευρώπη από τον επαναπατρισμό των ψηφιακών υπηρεσιών. Το εμπόδιο σε αυτό είναι η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων. Μέχρι το 2020 η Ευρώπη μπορεί να βρεθεί με έλλειψη 800.000 εργαζομένων στη ψηφιακή τεχνολογία. Δεν θα υπάρχουν αρκετοί νέοι. Τι κάνουμε λοιπόν για τη συγκεκριμένη ε, αγορά. Γιατί αυτή είναι πολύ σημαντική για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και Γιώργο Μπαλάς. Ευχαριστώ. Αυτές οι εισηγήσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Εγώ αυτό που με προβληματίζει είναι το εξή. Αν κατάλαβα καλά, θα μπορούσε να υπάρξει η επαναπατρισμός λόγω της αύξησης του κόστους εργασίας στην Κίνα ήταν πράγματα που έχουν συζητηθεί πριν από καμιά δεκαριά χρόνια. Ότι δηλαδή τη στιγμή που θα αυξηθούν οι μισθοί στην Κίνα, τότε θα γίνουμε λίγο περισσότερο ανταγωνιστικοί. Το πρόβλημα όμως είναι ότι εντωμεταξύ στην Ευρώπη, εκτός από το να προσπαθούμε να μειώνουμε κάπως τα ε, κοινωνικές προδιαγραφές, δεν έχουμε κάνει τίποτα παραπάνω όσον αφορά τις επενδύσεις, γιατί αν δει κανείς τι δυνατότητες της Ευρώπης να φτιάχνει προϊόντα και αντικείμενα νέα σε σύγκριση με αναδυόμενες χώρες αλλά και με τη ΣΥΠΑ, όχι μόνο η αδυναμία μας διαπιστώνεται, αλλά έχουμε μείνει πραγματικά πίσω σε αυτά τα θέματα. Και διαπιστώνουμε μάλιστα ταυτόχρονα μια μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων αλλά και μείωση των δημοσίων επενδύσεων. Διότι εφόσον έχουμε μεγάλη χρέωση, η εν δεν είναι για να γίνουν επενδύσεις αλλά για άλλους λόγους που συνδέονται με πολιτικές ε, παλιές αλλά και με την κρίση του 2008. Το ερώτημα λοιπόν που ήθελα να θέσω αφορά αυτές τις επενδύσεις σήμερα. Πώς λοιπόν οι επιχειρήσεις ε, αντιλαμβάνονται αυτό το θέμα. Στη Γαλλία περιμένουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις αλλά με το σταγονόμετρο έρχονται Ποια είναι το βασικό θέμα και αν μας πείτε πάλι είναι το κόστος της εργασίας το πρόβλημα, να σας πω δύο. Το κόστος εργασίας έχει μειωθεί. Το ρίο κόστος στη βιομηχανία είναι χαμηλότερο από ό,τι στη Γερμανία, αλλά αυτό δεν σημαίνει περισσότερες επενδύσεις, δεν έχουν έρθει περισσότεροι επενδυτές. Τώρα, αν μειωθεί ακόμα περισσότερο η ζήτηση, θα σημαίνει αυτό ιδιωτική χρέωση που ήταν το αίτιο της κρίσης του 2008. Γιατί έτσι είχε τη είχαν τη σταθμίσει, είπα, την τελμάτωση των μισθών για 30 χρόνια με ιδιωτική χρέωση. Πώς λοιπόν θα εμείς θα ελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σιμαρτά. Ευχαριστώ. Επιστροφή σημαίνει πρώτα αναχώρηση. Αυτό το είχαμε καταδικάσει, είχαμε προτείνει εθνικά μέτρα, αλλά δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά μέτρα. Επαναπατρισμός λοιπόν σημαίνει ποιοτική και ποσοτική μείωση της ανεργίας. Κάτι που δεν συμβαίνει από ό,τι βλέπω. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, αυτό δεν προκύπτει από μία ανάπτυξη στην Ευρώπη, αλλά από την ε, διακοπή της ανάπτυξης σε άλλες χώρες, Κίνα, Μπρίξ Είναι συγκυριακό λοιπόν και εξαρτάται από άλλες εξελίξεις της αγοράς στον κόσμο. Κατά την άποψή μας, αυτό μπορεί να, δεν μπορεί να γίνει με μια άκαμπτη υπερεθνική ευρωπαϊκή στρατηγική που αγνοεί τις ε, ε, ιδιαιτερότητες των χωρών. Άρα το ερώτημα που τίθεται είναι πού θα γίνει και πότε αυτή, αυτός ο επαναπατρισμός. Δηλαδή επιστρέφουν αλλά ίσως όχι στη χώρα προέλευση, σε μια άλλη χώρα της ευρωπαϊκής κοινότητας low cost. Τι αντίκτυπο θα έχει όμως κάτι τέτοιο. Θα οδηγούσε εν τέλει στο να έχει ένωση ε, θα μπορούσε να γίνει μόνο αν η Ένωση είχε πραγματικές αρμοδιότητες στον τομέα της απασχόλησης. Δεν προβλέπω κάτι τέτοιο. Εμείς αντίθετα φοβόμαστε ότι αυτή η επιστροφή έχει καθαρά οικονομικούς ε, τροτούς λόγους. Αυτή η απόφαση προκύπτει ενδεχομένως από την αύξηση της παραγωγής στην Κίνα ή της παραγωγής ε, της μεταφοράς από την Ασία και από την έλλειψη αντικαταστάτη της Κίνας. Αν εμφανιστεί ένα νέο Ελντοράντο θα ξαναφύγουν οι επιχειρήσεις απολύνοντας εκ νέου χιλιάδες άτομα. Αρχέτυπο αυτής της παγκοσμιοποίησης είναι ο κ. Καλντέιρα που πήγε να φάει το, μέλι στην Κίνα δεν είδε, έφαγε mail, μέλι, μετά τελείωσε το μέλι στην Κίνα, ήρθε στην Μεγάλη Βρετανία και έκανε και μια νέα κυψέλη στι Ηνωμένε Πολιτείε. Άρα δεν προστατεύει ούτε τα συμφέροντα τη Ευρώπη ούτε τα συμφέροντα τη Βρετανία. Τα δικά του κυνηγάει. Και μα λέει ότι είναι υπέρ της κατάργησης όλων των κριτηρίων, ε, της κατάργησης όλων των εμποδίων που θα του επιτρέψουν να ξαναφέρει αυτό το, αυτή την αμερικανική κυψέλη που έχει στη Βρετανία. Αλλά αυτό θα οδηγήσει σε είσοδο εκατοντάδων άλλων αμερικανικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και απολύσεις. Δεν μου προσέφερε κάτι η άποψη του κύριου Καλντέρια. Ο κύριος Καλντέρια υποστηρίζει τα συμφέροντά του τελεία και παύλα. Επίσης, η Επιτροπή έκανε ανάλυση, μελέτη, ανάλυση, ανάλυση αντικτύπου για να δει πού γίνονται αυτές οι επιστροφές. Ποιοι είναι οι τομείς και οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται. Ελπίζω ότι η ακρόαση θα βοηθήσει να καλύψουμε τις ενσυχίες μας και να τεκμηριώσουμε την προσέγγιση αυτή. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις. Προτείνω να ξεκινήσουμε με την ίδια σειρά. Κύριε Τόρες, Καλντέιδα, και μετά ο κύριος Σαλγκάδο. Τόρες. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Τι σημαίνει ανταγωνιστικότητα. Νομίζω ότι για χρόνια η ανταγωνιστικότητα αντιμετωπιζόταν μόνο ως κόστος. Ανταγωνιστικότητα όμω είναι η ικανότητα των οικονομιών της Ευρώπης να προσαρμοστούν και να αλλάξουν για να αντιδράσουν στις ε, μεγάλες αλλαγές τεχνολογίας και της οικονομίας. Αυτό είναι διαφορετικό από την ε, ανταγωνιστικότητα μόνο κόστου, λόγω κόστους. Αυτό γινόταν στο παρελθόν, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι το κόστος της νέας τεχνολογίας, αυτή η διαδικασία κατακαιρματισμού της παραγωγής που έγινε, οδήγησε αλλαγή των βασικών αξιών της οικονομίας. Η βελτίωση της νομοθεσίας λοιπόν είναι αναγκαία. Δεν θέλει λιγότερη ρύθμιση, αλλά προσαρμογή των ρυθμιστικών πολιτικών σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αυτό είναι σημαντικό. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ερώτηση τι εννοούμε με τον όρο better regulation, καλύτερη νομοθεσία. Σε εθνικό επίπεδο, τρεις είναι οι βασικές αρχές που είναι σημαντικές. Πρώτον, προστασία αυτών που πρέπει να προστατευθούν. Η Ευρώπη, νομίζω, για πολλά χρόνια λειτουργήσε καλά προστατεύοντας επιχειρήσεις, ανθρώπους και διεργασίες. Διότι μπορείτε να δείτε ότι σε πολλές περιοχές του κόσμου δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής νομοθεσίας που προστατεύει. Και αυτό περιλαμβάνει μονοπόλια και ανισότητες. Πρώτο λοιπόν στοιχείο η προστασία. Δεύτερον στοιχείο προβλεψιμότητα. Για όλους τους εργαζόμενους επιχειρήσει στην κυβέρνηση και σε κάποιες χώρες ε, η νομοθετική ρύθμιση είναι σύνθετη. Άρα το να είναι προβλέψιμη είναι πολύ σημαντικό. Τρίτον, να μην μπερδεύουμε τα δικαιώματα με τους κανόνες. Φερβίν στον τομέα της υγείας ή της συνταξιοδότησης, το δικαίωμα προστασίας της υγείας ή της, το δικαίωμα σύνταξη πρέπει να ε, το θέμα που τίθεται είναι ποιοι είναι οι κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων αυτών με, τους νέους, με τις νέες συνθήκες. Στην περίπτωση της Ελλάδας κάναμε μία μελέτη των μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας μετά την Κρήτη η πλειοψηφία πηγαίνει στην λιγότερη νομοθεσία, χωρίς αυτό να το κάνουμε. Χωρίς να το κάνουμε αυτό με καλύτερο. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να λάβουμε υπόψη αυτούς τους βασικούς κανόνες. Τώρα, υπήρχε μια ερώτηση για την καλύτερη νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το TTIP. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός, ε, το Παγκόσμιο Γραφείο Εργασία δεν έχει θέση για το TTIP, πρέπει να δει το τελικό κείμενο. Υπάρχουν ωστόσο εδώ κάποιε γενικές αρχές, μία από τις οποίες είναι ότι είναι σημαντικό ο εταίρος που έχει τους πιο προστατευτικούς κανόνες να είναι αυτός στον οποίο όπου θα υπερισχύει, του οποίου η νομοθεσία δεν υπερισχύει. Για παράδειγμα, οι βασικές συμβάσεις του Παγκόσμιου Γραφείου Εργασία έχουν επικυρωθεί από όλα τα κράτη της Ένωσης. Αυτό είναι πλεονέκτημα για την Ένωση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν κυρώσει και τις οκτώ συμβάσεις, βασικές συμβάσεις του ΠΟΕ στη διαδικασία αυτή εσείς έχετε λόγο για να παροτρύνετε τις είπα να σταθούν στο ίδιο επίπεδο με εσά. Το δεύτερο έχει να κάνει με την προστασία των επενδύσεων. Εδώ υπάρχουν δύο προβλήματα. Ο κίνδυνος ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών νομοθετικής και κανονιστικής ρύθμισης και εδώ ήταν χρήσιμο να υπάρχει αναφορά στο κείμενο ως προς το γεγονός ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοινωνική ή περιβαλλοντική νομοθεσία την προστασία της, ε, των επενδύσεων. Το άλλο έχει να κάνει με το ποιο αποφασι... ποιος αποφασίζει, ποιο δικαστήριο αποφασίζει σε περίπτωση που υπάρξει μια διαφορά. Στην Ευρώπη άκουσα μια ενδιαφέρουσα ε, πρωτοβουλία της δημιουργίας ενός οργάνου δημοσίου που θα κάνει αυτή την δραστηριότητα. Και κάτι άλλο. Γιατί διαφέρει η Ελλάδα σε σχέση με άλλους. Σε σχέση τώρα της Ευρώπης από τις χώρες των BRICS και θα έλεγα ότι η μεγάλη διαφορά της Ευρώπης είναι η μεγάλη μεσαία που έχει ε, γιατί παρέχει την ε, σταθερότητα στα εθνικά κοινοβούλια επιτρέποντας σε όλους να καταλάβουν ότι η πολιτική δουλεύουν για αυτούς και τα παιδιά τους. Η σταθερότητα και η δυναμική της μεσαίας τάξης λοιπόν είναι σημαντικό. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι νομίζω φορούσε τις αγορές εργασίας αυτό το ερώτημα, ότι είναι μια αγορά εργασίας βάσει κανόνων και αυτό προϋποθέτει τον σεβασμό το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του κράτους δικαίου που διαφέρει από χώρα σε χώρα αλλά που προβλέπει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε την κατάσταση σε μια σειρά χωρών. Το θεσμικό πλαίσιο λοιπόν είναι σημαντικό και είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί αποδυναμώνονται όργανα που εξυπηρέτησαν την Ευρώπη πολύ επειδή χρησιμοποιούνται επιχειρήματα που δεν αποδεικνύονται. Υπήρχε και μία ερώτηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το είπε ο κύριος Καλτέρα νομίζω. Το χρηματοοικονομικό σύστημα στην Ευρώπη δεν είναι προσαρμοσμένο. Έχει αλλάξει η οικονομία και αυτό έχει επιπτώσεις και στο οικονομικό σύστημα. Ένας λόγος για τους οποίους ε, οι επενδύσεις δεν έχουν, δεν έχουν υπερβαστεί, είναι, υπερ, δεν έχουν ε, αυξηθεί είναι διότι ακριβώς ε, δεν είναι δυνατόν να προγραμματίσουμε το πλαίσιο αυτό. Αν βελτιώσουμε το χρηματοοικονομικό σύστημα, μπορούμε να βελτιώσουμε τις επενδύσεις. Το private banking, ας πούμε, στην Ευρώπη, που δεν είναι τραπεζικό σύστημα, ευημερούν στην Ευρώπη διότι το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα δεν προσαρμόστηκε στην νέα ανάγκη να μεταφέρει τις αποταμιεύσεις τις επενδύσεις είχε μια ενδιαφέρουσα εικόνα στην παρουσίασή του ο κ. Καλντέρα για τον τραπεζικό δανεισμό. Θα σταματήσω εδώ και ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σα Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Καλτέρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που ακούστηκαν, γιατί ακούστηκαν πολλές. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια. Ζητώ συγγνώμη εάν δεν τις προλάβω όλες. Προσπάθησα να τις καταγράψω όσο πιο γρήγορα μπορούσα να απαντήσω ότι συμφωνώ με τον κύριο Τόρες όσον αφορά τις παρατηρήσεις του. Η μικρή μου διαφωνία αφορά τον δικό μου τομέα, όπου το κόστος αυξάνεται πολύ πιο γρήγορα στην Κίνα από ό,τι φαίνεται από ε, τα μακροδεδομένα. Αυτό όμως το βλέπω ε, από τη δική μου πείρα. Μπορεί λοιπόν ε, οι θέσεις εργασίας να φτάσουν πολύ πιο γρήγορα στην Ευρώπη. Στον κύριο Καρσία Σαλκάδο να πω ότι το δικό μου ένστικτο μου λέει ότι Δυστυχώς έχουμε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα ανεργίας νέων στην Ισπανία. Θέλουμε να διασφαλίσουμε βιώσιμες θέσεις εργασίας, μακροπρόθεσμες. Δεν θέλουμε να έχουμε ανταγωνισμό προς τα κάτω. Αυτό δεν θα είναι καλή ιδέα για την Ευρώπη. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσετε. Το πρόβλημα είναι όμως ότι οι εργοδότες θέτουν τους όρους στην Ισπανία. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εξαιρετικό παράδειγμα του αντιθέτου όπου βλέπουμε αύξηση των ε, μισών και αποδοχών ε, κατά 3% τον χρόνο, κάτι που οφείλεται όχι στην ομοθεσία αλλά στον ανταγωνισμό εντός αγοράς εργασίας. Εάν κάποιος δεν είναι ικανοποιημένος ε, με τη δουλειά του, εάν ο εργαζόμενος μου δεν είναι, ε, ο υπάλληλος μου δεν είναι ικανοποιημένος, σηκώνεται και θα φεύγει και πάει αλλού. Έτσι λοιπόν δεν είναι απαραίτητη η νομοθεσία για να ε, ανεβάσει τον πύχη ε, και ο ανταγωνισμός μπορεί να το κάνει αυτό. Καταλαβαίνω βέβαια ότι κάθε χώρα βρίσκεται σε άλλο μέρος του οικονομικού κύκλου, κάτι λοιπόν που μπορεί να ευνοήσει τον Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να μην ωφελήσει άλλους, αλλά ε, νομίζω ότι ο ανταγωνισμός περισσότερο από την νομοθεσία θα μας οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο Εδουαρδ έχει δίκιο ότι χρειάζεται κίνητρα θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για επιχειρήσεις που θέλουν να επαναπατριστούν, ε, επιχειρήσεις σαν τη δική μου που κοντεύουν να φτάσουν στο σημείο καμπής και ετοιμάζονται να λάβουν την απόφαση επαναπατρισμού των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Θα πρέπει να έχουν την κυβέρνηση σε οποιοδήποτε επίπεδο με το μέρος τους, είτε πρόκειται για την ευρωπαϊκή, εθνική ή περιφερειακή. Εάν πρόκειται για ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας και δεν πρόκειται για θέσεις που ε, ανταγωνίζονται προς τα κάτω, νομίζω ότι αυτό θα ωφελήσει τους εργοδότες, ε, τους επιχειρηματίες σε όλη ε, την Ευρώπη. Συμφωνώ με αυτά που είπε η Άνθια. Αναζητούμε τη μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας ώστε να είναι πιο εύκολο για τις επιχειρήσεις να προσλάβουν πιο εύκολα ανθρώπους, ώστε να είναι και οι επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές. Τα παραδείγματα της Ισπανίας είναι υπερβολικά. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Καρσία Σαλγάδο ότι το να, προσλάβει, το να προσλαμβάνει ε, κάποιος ανθρώπους τη Δευτέρα και να τους απολύει την Παρασκευή είναι γελίο. Εγώ ως ε, Βρετανός επιχειρηματίας δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν συμφωνούμε με τις βραχυπρόθεσμες ε, συμβάσεις εργασίας, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες. Όσον αφορά το θεματολόγιο για την καλύτερη νομοθεσία, η Ευρώπη θα πρέπει να καταλάβει ότι οι επιχειρήσεις και ε, οι επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο έχουν την επιλογή, μπορούν να επενδύσουν όπου θέλουν. Θα πρέπει λοιπόν η δική μας δουλειά, η δουλειά όσων βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, είναι να κάνουν την Ευρώπη όσο γίνεται πιο ελκυστική για επενδύσεις κεφαλαίων, αλλά και επενδύσεις ε, στην εκπαίδευση και τις δεξιότητε των ανθρώπων. Πιστεύω λοιπόν με όλο το σεβασμό ότι η δουλειά σας εδώ είναι ε, να κάνετε κάθε χώρα ξεχωριστά και την Ευρώπη στο σύνολό της όσο γίνεται πιο ελκυστική για τους επενδυτές. Αυτό γενικά σημαίνει καλύτερη νομοθεσία, όχι απαραίτητα έλλειψη νομοθεσίας, ε, απορρίθμιση, αλλά καλύτερη νομοθεσία και περισσότερο ανταγωνισμό. Κυρία Στάινρουκ. Έχετε δίκιο. Η αγορά είναι παγκόσμια, ο ανταγωνισμός είναι παγκόσμιος. Εγώ ο Καλτέρα ανταγωνίζομαι σε παγκόσμιο επίπεδο όπως και η Ευρώπη. εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό είναι απαραίτητο. Νομίζω ότι η ιδέα του να, χρησιμοποιηθούν, το να χρησιμοποιηθεί φορολογία των επιχειρήσεων ε, στις υποδομές που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις αυτές είναι λογική ιδέα, αρκεί να μην είναι τόσο απαγορευτική φορολογία που οι επιχειρήσεις αυτές ε, να μην μπορούν να έχουν κέρδος και να επενδύουν και μόνες τους. Είναι σημαντικό σαν, ως να έχουμε την ε, σωστή υποδομή, να έχουμε μακροπρόθεσμες επενδύσεις, να επαναπατρίσουμε τις επιχειρήσεις, όχι όμως να τις φορολογούμε σε βαθμό που να μην είναι πια ανταγωνιστικές και που να μην είναι πια ανταγωνιστική η πυρός μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φράση σας ότι τα αυτοκίνητα δεν πολλούν αυτοκίνητα και η απάντηση εδώ είναι ο ανταγωνισμός. Όσον αφορά την ε, ερώτηση που θέσατε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ξύσαμε το εργατικό μας δυναμικό κατά 20% και μειώσαμε το κινέζικο εργατικό δυναμικό κατά 25%. Πήραμε λοιπόν τις θέσεις εργασίας που είχαν μετεκατασταθεί στην Κίνα και τις φέραμε πίσω αλλά η δουλειά μας είναι κάπως πιο δύσκολη τώρα, διότι τώρα είμαστε έτσι μια διεθνής επιχείρηση. Όσον αφορά την ερώτηση της Μαριαρένα, έχει δίκιο. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι κατακαιρματισμένη η παγκόσμια οικονομία, είναι πολύπλοκη και μόνο οι επιχειρήσεις και οι χώρες που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της κατακαιρματισμένης παγκόσμιας οικονομίας θα επιβιώσουν ο Υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου χρησιμοποιεί μια έκφραση που έκλεψε από έναν πολιτικό που βοήθησε στην ανοικοδόμηση του Λίβερπουλ τη δεκαετία του 1980. Είπε ότι συμμετέχουμε σε έναν παγκόσμιο αγώνα ε, ως μεμονωμένες χώρες και ως ε, μεμονωμένες επιχειρήσεις. Όσον αφορά την συμφωνία TTIP, η δική μου προοπτική είναι πολύ απλή. Η Καλτέρα ε, ε, έχει ε, είναι διεθνής επιχείρηση, πολλούμε και αγοράζουμε στην παγκόσμια αγορά. Με μείωση των δασμών στις ΗΠΑ θα έχουμε τη δυνατότητα να αγοράζουμε τα προϊόντα μας από την ε, Ευρώπη, αγοράζουμε υφάσματα στην, ε, στο Βέλγιο, στην Ιταλία, στην Ισπανία, κατασκευάζουμε τα προϊόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε λοιπόν θέσεις απασχόλησης, ε, στηρίζουμε θέσεις απασχόλησης και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο υπόλοιπο της Ευρώπης, πολλούμε τα προϊόντα αυτά στις Ηνωμένε Πολιτείες, και αυτέ είναι θέσει απασχόληση που πριν βρίσκονταν στην Κίνα. Τώρα δηλαδή αντικαθιστούμε τα προϊόντα που προέρχονταν από την Άπο Ανατολή ε, με προϊόντα ε, που κατασκευάζονται τώρα πια στην Ευρώπη. Επίσης, μου τέθηκε η ερώτηση για τον ΠΟΕ και την μετεκατάσταση της καλτέρα στην Κίνα. Η επιχείρησή μας έπρεπε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετώπιζε. Ε, μπορεί κανείς να αντιδράσει με διαφορετικούς τρόπους, αλλά οι πιο ακραίες ε, αντιδράσεις θα ήταν ή να αντιδράσει ή να αγνοήσει τις προκλήσεις. Ε, υπήρχαν πολλές εταιρείες που χρεοκόπησαν και χάθηκαν όλες οι θέσεις εργασίας. Εμείς ως αμυντική κίνηση πήγαμε στην Κίνα, διότι οι άνθρωποι που έχουν επιλογή σχετικά με το από πού θα αγοράσουν προϊόντα ήθελαν προϊόντα βρετανικά αλλά με κόστος κινέζικο. Έτσι λοιπόν ε, μεταφερθήκαμε στην Κίνα ε, για να μειώσουμε το κόστος. Αλλά αυτό που συνέβη ήταν ε, περίεργο διότι συμμετείχαμε σε εκθέσεις στην Κίνα με προϊόντα βρετανικού σχεδιασμού κατασκευασμένα στην Κίνα. Διπλασιάστηκα η επιχείρησή μας τα πρώτα δύο χρόνια και μετά ξαναδιπλασιάστηκε τα επόμενα δύο χρόνια διότι πολλοί άνθρωποι βρήκαν εξαιρετικό συνδυασμό ευρωπαϊκού σχεδιασμού και κινέζικης παραγωγής. Έτσι, ε, προστατεύσαμε κάποιες θέσεις απασχόλησης ε, στον σχεδιασμό, στην, ε, στο τμήμα πολίσεων, στο οικονομικό τμήμα και έτσι όχι μόνο σώθηκε η επιχείρησή μας, διότι όπως ανέφερα κλείσαμε το ένα μας εργαστήριο, αλλά διατηρήσαμε ένα από τα εργοστάσια μας. Αλλά επειδή καταφέραμε να αντιδράσουμε, δημιουργήσαμε και μια παγκόσμια ευκαιρία. Μετατρέψαμε μια απειλή σε ευκαιρία διότι στο παρελθόν δεν είχαμε τη δυνατότητα να πολλούμε σε χώρες όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι άλλες αναδυόμενες αγορές, διότι δεν μπορούσαμε να ανταγωνιζόμαστε τα ε, κινέζικα προϊόντα. Έτσι όμως γίναμε μια εταιρεία ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, ναι, ναι. Όσον αφορά τις Ηνωμένε Πολιτείε, ε, σκοπό είχαμε να ε, πολλούμε προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα, στις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά τώρα πολλούμε περισσότερα από τα προϊόντα μας που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε. Στο κατάστημά μας λοιπόν στην Νέα Υόρκη βλέπουμε ότι πολλούνται περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα και αφαιρούνται τα κινέζικα προϊόντα. Με τη συμφωνία TTIP θα έχουμε συνθήκε ίσου ανταγωνισμού. Είναι ήδη δύσκολο για εταιρείε παραγωγή τη Ευρώπη να πολλούν στι ΗΠΑ επειδή ε, ε μα εμποδίζει ο Ατλαντικό ωκεανό. Έχουμε λοιπόν κόστο μεταφορών. Εάν όμω αφαιρέσουμε του δασμού και έχουμε συνθήκε ίσου ανταγωνισμού, με ε, Βεβαίω ότι θα μπορέσουμε να εξωθήσουμε από την Αμερικανική αγορά ειδικά και Κινέζικα προϊόντα και θα μπορέσουμε να τα αντικαταστήσουμε με ε, προϊόντα κατασκευασμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό είναι ένα θετικό τρόπο να δούμε το TTIP. Να απαντήσω στην Μαρτίνα ότι είναι πολύ χρήσιμε οι εμπειρίε τη από τον πραγματικό κόσμο. Πιστεύω ότι ε, πρέπει περισσότεροι επιχειρηματίε να συμμετέχουν στην πολιτική, διότι αυτό ε, διευκολύνει την κατανόηση και μάλιστα την ε, παραγωγή πλούτου και όχι απλά την ανακατανομή πλούτου. Ο ανταγωνισμός είναι πραγματικότητα. Ε, αυτά δεν είναι πράγματα που, δεν θα πρέπει να, που θα πρέπει να αρνούμαστε να συζητήσουμε. Στην πραγματικότητα οι επιχειρήσει θα μετακατασταθούν εκεί που μπορούν να κερδίσουν περισσότερα. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, διότι τελικά, εάν δημιουργείται πλούτο, εάν δημιουργείται κέρδο, ε, όπω υπόθηκε πριν, δεν αγοράζουν τα αυτοκίνητα αυτοκίνητα, οι άνθρωποι αγοράζουν τα αυτοκίνητα. Ε, έτσι λοιπόν ε, θα είναι καλό αυτό. Η πρόσβαση στις ε, νέες αγορές μέσω ε, ε, του κινέζικου μας εγχειρήματος ήταν πολύ σημαντικό και αγορές που μας ανοίχθηκαν έτσι ε, εξυπηρετούνται τώρα με τα ευρωπαϊκά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν, επειδή αντιδράσαμε σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα, δημιουργήσαμε μία παγκόσμια επιχείρηση, μία παγκόσμια λύση. Αυτό λοιπόν αποτελεί ένα μικρό παράδειγμα του τι κάνει η επιχείρησή μου και νομίζω ότι είναι σημαντικό για τους πολιτικούς εδώ, διότι αυτό που θα πρέπει να καταφέρουμε εδώ μέσα είναι να εξετάσουμε την απειλή που αντιμετωπίζουμε και να την μετατρέψουμε σε ευκαιρία. Όσον αφορά τους νέους και την ερώτηση της ε, Μαρτίνα, είμαστε προορατικοί, δημιουργούμε νέα προϊόντα, έχουμε εξαιρετικούς σχεδιαστές στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε προϊόντα που σίγουρα δεν μπορούν να σχεδιαστούν στην Κίνα. Το ίδιο ισχύει στην Ευρώπη. Ακόμα και ο Κινέζος θα προτιμούσε ένα γερμανικό αυτοκίνητο και ένα ιταλικό κουστούμι αντί για κινέζικα. Η συζήτηση περί επαναπατρισμού λοιπόν ε, δεν είναι, είναι πολύ σημαντική όχι μόνο όσον αφορά τις ε, θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη αλλά πρέπει να θυμόμαστε και τον ρόλο της μεσαίας τάξης στην Κίνα. Έχουμε την ευκαιρία να μετατρέψουμε μια αμυντική στρατηγική σε κερδοφόρο στρατηγική για την Ευρώπη. Η αναδυόμενη μεσαία τάξη στην Κίνα ε, δεν θα γίνει η παραγωγή, θα γίνει οι καταναλωτές. Και επιχειρήσεις σαν τη δική μου ε, προσλέπουν στις, ε, στην αύξηση των πωλήσεων προς την Κίνα. Όταν πρωτοπήγαμε στην Κίνα πριν 10-12 χρόνια, αν μου λέγατε ότι σε 10 χρόνια θα επαναφέρουμε θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και θα πολλούμε προϊόντα στην Κίνα, εγώ θα του έθελα στον ψυχίατρο, διότι πίστευα ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ποτέ. Αλλά σήμερα αυτό ακριβώς βλέπουμε. Και άλλη μια πολύ καλή ερώτηση από την Μαρτίνα για την ψηφιακή οικονομία. Έχουμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα αυτόν τον μήνα, στις αρχές του μήνα, στις Βρυξέλλες, στο κέντρο Expo, είχαμε μια έκθεση που λεγόταν Mood ε, στον τομέα των υφασμάτων. Είναι πολύ σημαντική εκδήλωση αυτή ε, για τους ανθρώπους στον τομέα των υφασμάτων. Ε, με φέρνει τακτικά στις Βρυξέλλες και αγαπώ πολύ την πόλη αυτή. Φέτος βρήκαμε μια ισπανική εταιρεία που είχε επενδύσει πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, μικρομεσαία επιχείρηση, που είχε επενδύσει σε ε, ψηφιακά μηχανήματα εκτύπωσης. Ε, ε, βρήκαν λοιπόν έναν τρόπο να κατασκευάσουν το προϊόν πιο φθηνά από τους Κινέζους ανταγωνιστές τους. Μέσα στο τελευταίο μήνα μόλις, μια ισπανική εταιρεία επένδυσε σε ψηφιακή τεχνολογία εξωθώντας τα κινέζικα προϊόντα και επαναφέροντας θέσεις εργασίας. Και τώρα έχουν προσλάβει πολιτές, σχεδιαστές και ενώ πριν είχαμε ε, υφάσματα εμπριμέ από την Κίνα, τώρα έχουμε υφάσματα εμπριμέ από τη Βαλένθια. Βλέπουμε λοιπόν εκεί αύξηση των θέσεων απασχόλησης, ε, αύξηση των δραστηριοτήτων που βασίζεται σε προώθηση μιας ψηφιακής τεχνολογίας. Ακόμα λοιπόν και στον ταπεινό τομέα των υφασμάτων βλέπουμε την ψηφιακή επανάσταση. Και να κλείσω με την ερώτηση του Γκί. Είναι σημαντικό οι πολίτες να καταλάβουν ποιο είναι το σημείο κάμπης για κάθε επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση πρέπει να λάβει μια απόφαση πότε θα επαναπατρίσουμε τις ε, εγκαταστάσεις μας. Εάν λοιπόν ε, τα δίκτυα υποστήριξη των επιχειρήσεων μπορούν να το καταλάβουν αυτό, ε, θα μπορέσουν να συνεργαστούν με τους ε, πιθανούς εργοδότες για να επιταχύνουν τη διαδικασία αυτή, διότι η διαδικασία αυτή ε, θα φέρει όχι μόνο θέσεις απασχόλησης άμεσες, αλλά και θέσεις απασχόλησης μέσω της αλυσίδας προμήθειάς τους. Στην πόλη μου έχουμε το εργοστάσιο της Vauxhall, έχουμε την τύχη αυτή βλέπουμε ότι είναι τεράστιο πλεονέκτημα να παράγονται περισσότερα προϊόντα σε μια οικονομία. Και όσον αφορά την προοπτική των επενδύσεων. Ο σχεδιασμός, η προστιθέμενη αξία, η δημιουργική διαδικασία. Η Ευρώπη είναι η πιο δημιουργική ήπειρος σε όλο τον κόσμο. Έχει ιδέες, καινοτομία, ηγείται στους τομείς αυτούς και είμαι πολύ περήφανος που το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια από τις καινοτόμες αυτές χώρες. Με τη δημιουργία νέων προϊόντων, νέων ιδεών έχουμε την δυνατότητα να φέρουμε τα προϊόντα μας στο, στην παγκόσμια σκηνή και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες σε διεθνές επίπεδο. Όσον αφορά την επίκριση του Ντομινίκ, ε, καταλαβαίνετε ότι θα διαφωνήσω με τα περισσότερα πόσα όσα υπόθηκαν. Σημαντικό είναι όχι μόνο ο Ντομινίκ, αλλά και άλλοι να μην θέτουν ε, την ερώτηση ρωτώντας ε, αν, αλλά εγώ είμαι η ζωντανή απόδειξη ότι θα πρέπει να ρωτάνε πότε θα γίνει αυτό. βλέπετε ότι οι άμεσες ε, ξένες επενδύσεις, ε, ότι έχουμε ε, μεταστροφή στον τομέα των άμεσων επενδύσεων προς όφελος της Ευρώπης. Πέρα λοιπόν από το δικό μου ταπεινό μικρό παράδειγμα μπορούμε να δούμε και άλλα παραδείγματα σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αυτά είναι καλύτερα θα είναι καλά νέα για την ε, Ήπειρό μα Ας αδράξουμε την ευκαιρία. οι επιχειρήσει ε, μετακαταστάθηκαν για ε, οικονομικού λόγου. Αυτή είναι η δουλειά των επιχειρήσεων, δημιουργούν πλούτο. Και μετά υπάρχει βέβαια το θέμα της ανακατανομής του πλούτου που δημιουργείται και υπάρχουν διάφοροι τρόποι να γίνει αυτό. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, αλλά επί της αρχής ε, αυτό ισχύει. Και όσον αφορά την κατηγορία ότι ο κύριος Καλτέρα απλά δοκιμάζει την τύχη του οπουδήποτε και ε, σκέφτεται μόνο το χρήμα. Να σας πω ότι η επιχείρησή μας ε, μίκρινε ε, κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ε, διατήρησε όμως το ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό, ε, διατήρησε τους ευρωπαϊκούς προμηθευτές και χάρη σε αυτό τώρα αναπτύσσεται. Κλείνοντας, Θα ήθελα να πω ότι η επιχείρηση Καλτέρα ε, πέτυχε σε παγκόσμιο επίπεδο επειδή είναι ε, σε παγκόσμιο επίπεδο ανταγωνιστική και αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα του τι θα πρέπει να κάνει η Ήπειρος ε, συνολικά. Η Ευρώπη θα πετύχει εάν είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορεί να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε προταξιονιστικά μέτρα αλλά θα πετύχουμε μόνο εάν είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε μεταρρυθμίσεις και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Η επιχείρηση Καλτέρα ε, ε, επιβίωσε και τώρα είναι ανταγωνιστική. Και το μάθημα που μπορεί να μάθει η Ευρώπη από αυτό είναι ακριβώς το ίδιο. Εάν μπορέσουμε να μάθουμε, να προσαρμοστούμε, να μεταρρυθμιστούμε, να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί ως Ήπειρος, όχι μόνο θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε, αλλά θα αναπτυχθούμε και πάλι και θα ε, κατέχουμε ηγετική θέση στον κόσμο. Αυτό ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε. ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Σύντομη ερώτηση και σύντομη απάντηση παρακαλώ. Μία σύντομη υπενθύμηση. Σας ρώτησα εάν έχετε εμπειρίες, κύριε Καλτέρα. Εάν γνωρίζετε πολλές άλλες επιχειρήσεις που ε, ε, επανέφεραν θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Okay. In 2012... Ναι, το 2012 η εταιρεία επελέγει από το BBC, το εθνικό μας τηλεοπτικό σταθμό, για να κάνει ε, μια, ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται Town Taking στην Κίνα. Ήταν η ιστορία της ε, εταιρεία μας και πώς χρειάστηκε να μικρύνουμε στην ε, Κίνα και να μετά να επαναπατριστούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και ακολουθούσε τα εμπορικά επιχειρήματα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο γίνανε όλα αυτά. Υπάρχει στο YouTube αν θέλετε να το δείτε. Αυτό που ήταν ε, συναρπαστικό στη διάρκεια αυτού του ντοκιμαντέρ ήταν ο αριθμό των άλλων εταιριών που προσπαθούσαν να κάνουν ακριβώ το ίδιο πράγμα. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που μέχρι ότου να ολοκληρωθεί το ντοκιμαντέρ η παραγωγή είχαν λάβει εκατοντάδε πληροφορίε, αλλά και αιτήματα από άλλε εταιρείε που ήθελαν να συμμετέχουν στο ντοκιμαντέρ. Αυτό ήταν το 2012, όχι 2015. εκατοντάδε και ίσω και χιλιάδε ε, επιχειρήσει σε ολόκληρη την Ήπειρο που προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Δεν είμαστε εμείς οι πρωτοπόροι, ε, δεν είμαστε μόνοι μας. Ναι, ε, είμαστε από τους πρώτους, αλλά είμαστε βέβαιοι ε, και μετά από αυτό το ντοκιμαντέρ ότι πάρα πολλές ακόμα εταιρείε κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σαλγάδο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομο. Θέλω να πάω και Βαρκελόνη, δεν θέλω να αργήσω. Νομίζω ότι δεν υπάρχει σωστός ορισμός για το τι σημαίνει ανταγωνιστικότητα. Ε, έχω, πρέπει να έχουμε κανόνες παιχνιδιού και με αυτούς τους κανόνες να προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μία ανταγωνιστικότητα. Αλλά με ποιο μοντέλο, με μοντέλο πείνας ή με το μοντέλο που έχουμε. Ε, το ότι οποιαδήποτε γάτα σκοτώνει ποντίκια δεν μπορεί να είναι μια πολιτική της Ένωσης. Τώρα, ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης. Ποιότητα, δημοκρατία, σχέδιο, ε, τα διπλώματα, καταχωρημένα ε, διπλώματα τεχνίας, μέτρα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θυσιάζονται ε, ή που, δεν, που χάνονται γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση στην ε, τραπεζική, στον τραπεζικό δανεισμό και αυτό είναι μια λυσίδα γιατί όταν αποτυγχάνουν ή κλείνουν μικρές επιχειρήσεις αφήνουν πίσω τους καμένη γη που δύσκολα μπορεί να ανακτηθεί. Σε... Εγώ έρχομαι από μια χώρα όπου το 90% της βιομηχανίας γίνεται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από ανθρώπους που πίστευαν ότι έπρεπε να επενδύσουν τα χρήματα και τις γνώσεις τους στην παραγωγική οικονομία και όχι στην κερδοσκοπία. Κάτι αξιοπρεπές, σημαντικό. Πρόσβαση λοιπόν στη χρηματοδότηση έργων που βελτιώνουν τις υποδομές πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές μας ε, στην Ευρώπη όχι μόνο γιατί χρειαζόμαστε και πρέπει να, να, να ανακαινήσουμε παλιέ. Ένα ενεργειακό πρόγραμμα για την Ευρώπη είναι αναγκαίο για την ανταγωνιστικότητα τη μελλοντική οικονομία και τη θέση εργασία που δημιουργεί η βιομηχανία και αποδεικνύει άλλωστε ότι είναι τομέα που μπορεί να δημιουργήσει θέσει εργασία ποιότητα. Η Ευρώπη χρειάζεται ένα ενεργειακό μοντέλο που συνδέεται απόλυτα με την ανταγωνιστικότητά τη και την πρόοδό τη τομείς που στην Ισπανία λειτουργούν καλά αυτόν τον καιρό είναι ακριβώς εκεί όπου υπάρχει ισορροπία μεταξύ συλλογικού, συλλογικών διαπραγματεύσεων και κοινωνικού διαλόγου, τα αυτοκίνητα. Είμαστε ο δεύτερο αυτοκίνητο παραγωγό στην Ευρώπη και μάλιστα ο διάλογο είχε ξεκινήσει πριν από πέντε χρόνια. Διότι το να δημιουργηθεί ένα αυτοκίνητο καθυστερεί πέντε χρόνια από τότε που ξεκινάει ο προσχεδιασμό μέχρι το πρωτότυπο του οχήματο χώρος των, ε, της αεροναυπηγικής επίσης λειτουργήσε ε, καλά. Διαπιστώσαμε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργήσει με ευάλωτες θέσεις εργασίας, ε, απορρίθμιση, γιατί σε λίγα χρόνια οι μισθοί θα είναι ψηλοί στην Κίνα και ε, ευάλωτοι στην Ευρώπη η αβέβαιη θέση εργασίας ε, ενός ανθρώπου σημαίνει ότι ο άλλος δεν καταναλώνει, δεν αγοράζει, δεν ψωνίζει, δεν αγοράζει αυτοκίνητο κατά συνέπεια, μειώνει την οικονομική δραστηριότητα. Και να σας πω ότι με τα μέτρα είναι ψέμα ότι ε, μειώθηκαν οι ανισότητες στην Ισπανία με την μεταρρυθμίση της, της ε, εργασιακής νομοθεσίας. Αυτό που έκανε το τελευταίο κείμενο είναι η καταστροφή σχεδόν ενό εκατομμυρίου θέσεων εργασία στην Ισπανία, 800 τόσε χιλιάδε. Και για κάθε μία που καταστρέ, καμία θέση που χάνεται δημιουργούνται ε, τέσσερις θέσεις ε, ευάλωτων ε, ε, προσωρινών θέσεων εργασίας. Το μοντέλο που ακολουθείται στην Ισπανία είναι αποτυχημένο και η Ισπανία λειτουργεί ως εργαστήριο που θέλει να εφαρμοστεί στην Ευρώπη και ελπίζω να μην εφαρμοστεί γιατί είναι διαπιστωμένο ότι έχει αποτύχει. Πάντα υπάρχουν, θα υπάρχουν χώρες που παράγουν φθηνότερα, θα παράγουν φθηνότερα από την Ένωση. Τα άτομα δεν είναι υλικό αγοραπολισίας. Ίσως θα έπρεπε οι πολιτικοί να καταλάβουν καλύτερα γιατί γίνεται αν οι πολιτικοί απλά παρακολουθούν ε, τις εξελίξεις των ε, δημοσκοπήσεων, αυτό είναι επικίνδυνο. Η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας επηρέασε κώδικες και συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Ντροπή για τον Υπουργό Εργασίας στη χώρα μου. Ε, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ο άνθρωπος αυτός θα έπρεπε να γυρίσει σπίτι του τι κάνουν οι Ευρωπαϊκές Σύνοδοι Απασχόλησης. Τέλο πάντων, εμεί είχαμε κάνει διάφορες εκδηλώσει κατά τη μεταρρύθμισης Τι θέλω να πω. Μίλησα για τα προβλήματα. Εναλλακτικέ. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων ε, και Βιομηχάνων παρουσίασαν στο Κοινοβούλιο για το πώ πρέπει να ξαναβάλουμε την βιομηχανία να δουλεύει. Είναι μεγάλες, υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις. Καλή ψηφιακή θεματολογία, αλλά αν δεν ε, μετέχουν όλοι, ε, δεν θα προχωρήσει. Πρόκειται για κάτι σημαντικό διότι επιτρέπει, θα επιτρέψει στην Ευρώπη να ανταγωνιστεί τις αγορές της Ασίας με βάση σημαντικές αξίες, αυτές που ανέφερα. Και η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείες πρέπει να γίνει δεκτή από τους πολίτες, ε, να είναι πιο ανοιχτή, πιο διάφανη και να υπάρχουν κανόνες που επιτρέπουν στους πολίτες να αποδεχθούν αυτή τη νέα πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και τη συμβολή σας. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα με πολύ συγκεκριμένα θέματα και παραδείγματα. Ακριβώς επί των ζητημάτων που μας απασχολούν σε αυτή την Επιτροπή. Όλοι σας τα αναφέρατε. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ θερμότατα. Ελπίζω να έχετε μια καλή επιστροφή. Uh, Προχωράμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, μικροχρηματοδότηση για την κοινωνική ένταξη. Ανταλλαγή απόψεων για την ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα δώσω το λόγο καταρχήν στην κυρία Ιβάνοβα. Θα ακούσουμε την εισήγησή σας και μετά θα έχετε το λόγο για να υποβάλλετε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πάντοτε μεγάλη μου χαρά να έρχομαι στην Επιτροπή Απασχόληση. Θυμάμαι ακόμα την τελευταία μας συζήτηση για την έκθεση της ε, εγγύηση για την νεότητα, για την νεολαία. Ελπίζω ότι το ίδιο ενδιαφέρουσα συζήτηση θα γίνει και για την μικροχρηματοδότηση. Η ερώτηση βασική ήταν κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σωστά τις ανάγκες των μικροεπιχειρηματιών. Αυτή την έκθεση τη δημοσιεύσαμε πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα, την παρουσιάσαμε τη Δευτέρα στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού και σας ευχαριστώ σήμερα που βρίσκομαι εδώ. Να σας δώσω λίγες πληροφορίες για το θέμα και τη σημασία του. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι μικροεπιχειρηματίες παίζουν ένα κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση του αποκλεισμού από την αποσχόληση μέσω της δημιουργίας μικροεπιχειρήσεων και νεοφυών επιχειρήσεων. Ωστόσο, ξέρουμε πως εν γέννη ε, έχουν δυσκολίες ε, στην πρόσβαση στην ε, παραδοσιακή αγορά πίστοσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να προσφέρει λύσεις. Η οικονομική στήριξη που προσφέρεται βασικά προσφέρεται μέσω του Κοινωνικού Ταμείου. Για την περίοδο μέχρι το 2013 είχαμε χορηγήσει συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω δανείων ή εγγύησεων ή και εγγύησεων. Άλλη σημαντική πηγή είναι το EPMF, το, η διευκόλυνση για την πρόοδο εξ ονόματος είναι ένα επενδυτικό ταμείο και διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω δανείων ή και εγγύσεων. 96 από τα 117 επιχειρησιακά προγράμματα του ESF για την περίοδο 2007 μέχρι 2013 χρηματοδότησαν τα μέσα υπό το τίτλο στήριξη για την αυτοαποσχόληση. Πρόκειται κυρίως για επιχορηγήσεις που ανήλθαν γύρω στα 2,4 δις ευρώ. Σε μικροεπιχειρηματίες, μάλλον το, το ακριβές ποσό που κατευθύνθηκε στους μικροεπιχειρηματίες δεν είναι γνωστό. Μέχρι το 2013 είχαν δοθεί 680 εκατομμύρια ε, ενώ το EPMF 203 εκατομμύρια ευρώ είχε δώσει για την περίοδο 2010 ε, μέχρι το 2013 και τα 103 από αυτά ήταν από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Όπως ξέρετε πρόκειται για μεγάλα ποσά, όπως βλέπετε μάλλον πρόκειται για μεγάλα ποσά. Προσπαθούμε να αναλύσουμε καλύτερα και να δούμε και πόσο αποτελεσματικά ήταν, αποτελεσματική ήταν αυτή η χρηματοδότηση. Θέλαμε λοιπόν να εκτιμήσουμε κατά πόσο οι ανάγκες των μικροεπιχειρηματιών καλύπτονταν από το ESF e, e και το EPMF. Πέντε κρατημέλη, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Ρουμανία εξετάστηκαν για να δούμε κατά πόσο η χρηματοδότηση αυτή επέτυχε στην παροχή χρηματοδότηση στους μικροεπιχειρηματίες. Επίσης, συγκεντρώσαμε τις διαθέσιμες πληροφορίες από τα κρατημέλη και την Κομισιόν σε σχέση με τα κόστη εφαρμογής. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το κόστος εφαρμογής είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και πάλι βρήκαμε αδυναμίες, αλλά πιστεύω πως είναι και χρήσιμο να τις τονίσουμε αυτές τις αδυναμίες, γιατί μπορούμε έτσι να αποκομίσουμε ε, διδάγματα, να βγάλουμε συμπεράσματα και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τις δυσκολίες αυτές στο μέλλον. Εν γέννη βρήκαμε αδυναμίες στον προγραμματισμό και το σχεδιασμό. γιατί δεν είχε γίνει ε, πάντοτε κατάλληλη αξιολόγηση των αναγκών Επίσης είχαμε κατάλληλα συστήματα διαχείρισης κινδύνου. Δεν είχαμε εξάλλου και αξιόπιστα στοιχεία όσον αφορά την απόδοση, γιατί ήταν έτσι δυνατό, αδύνατο να φτάσουμε σε ένα συνολικό συμπέρασμα σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των κονδυλίων που δόθηκαν στους μικρο, ε, μικρο, μικρο μάλλον, επιχειρηματίες. Εν γέννη όμως μπορούσαμε να πούμε ότι οι μικροεπιχειρηματίες ε, μπόρεσαν να πάρουν χρηματοδότηση. Μισή από αυτούς ήταν άνεργοι προηγούμενα και έτσι το πρόγραμμα αυτό ανταποκρίθηκε στις ανάγκες τους. Γενικό συμπέρασμα ήταν ότι καλύτερα αποτελέσματα θα είχαμε αν είχαμε αξιολογήσει καλύτερα και κατάλληλα τις ανάγκες τους, τις ειδικές τους ανάγκες, με βάση Έχουμε συντάξει κάποιες συστάσεις για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των διαθέσιμων κονδυλίων, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση συστήνουμε στα κρατημάλη να φτιάξουν ε, αξιολογήσεις όταν σχεδιάζουν τις ανάγκες και να ορίσουν επιχειρησιακά προγράμματα που περιλαμβάνουν την ε, ε, στήριξη στους μικροεπιχειρηματίες. Επίσης συστήνουμε στη Κομισιόν να χρησιμοποιήσουν τα στιβαρά συστήματα διαχείρισης κινδύνου. Επίσης συστήνουμε στη Κομισιόν και στα κράτη-μέλη να σχεδιάσουν μέτρα για να φτάσουν στις ευάλωτες ομάδες και στους ανέργους και τέλος τους συστήνουμε να αναλύσουν καλύτερα το κόστος εφαρμογής των διαφέρων επιδοτήσεων, πιστώσεων, δανείων, εγγύσεων, για να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και να μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες ε, ε, πρακτικές. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν σε καλύτερη οικονομική στήριξη στους μικρό επιχειρηματίες. Αυτά εν συντομία περιέχει η ε, έκθεση. Φυσικά θα περιμένω τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Και στρέφομαι στον κύριο Σούλτς που είναι ο εισηγητής. μπορείτε να προσθέσετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαρίστω. Θα προσπαθήσω αυτή τη φορά να τηρήσω και τον χρόνο ομιλία που μου δίνετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, εισαγωγική σας παρέμβαση. Διάβασα και όλο το κείμενο, 34 σελίδες ήταν το γερμανικό κείμενο, πρέπει όμως ε, να ομολογήσω ότι πολλά πράγματα δεν τα κατάλαβα κατά 100%. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ σήμερα να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχά ε, μου έκανε εντύπωση το ότι κάνετε εδώ μια σύγκριση ανάμεσα στο ESF που είναι ένα γενικό ταμείο και το πιο ειδικό ταμείο το EPMF το οποίο ε, έχει δημιουργηθεί ειδικά για την μικροχρηματοδότηση αλλά είναι σαν να συγκρίνουμε μήλα και πορτοκάλια. στα επιχειρησιακά προγράμματα υπήρχαν κάποια μέσα όπου υπάρχουν διαφορές. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε συγχρηματοδότηση στο ESF, ενώ στο EPMF έχουμε πιο πολύ εγγυήσεις και πιστώσεις. Εσείς βρίσκετε δηλαδή ότι είναι έγκυρη αυτή η σύγκριση. Έχω κάποιες αμφιβολίες. Πολύ ε, αξιέπαινο στην έκθεση βρήκα ότι ε, το κόστος ε, διαχείρισης του EPMF έρχεται σε 0,5 έως 1% ενώ στο ESF βρίσκεται στα 3,2%. Είναι αρκετά σημαντική αυτή η διαφορά. Έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Είπατε ότι εξετάσατε πέντε χώρες, μεταξύ άλλων την πατρίδα μου, τη Γερμανία. Η Γερμανία όμως ε, στο δεν συμμετέχει καν στο πρόγραμμα μικρό ε, πιστώσεων Progress. Ε, γιατί παρόλα αυτά εξετάσατε τη Γερμανία και μία ακόμα παρατήρηση, όχι ερώτηση ακριβώς, πιο πολύ παρατήρηση. Αν κατάλαβα καλά την έκθεση του ελεκτικού συναδρίου, μία συνέπεια είναι να αναλυφθεί το EPMF ε, από ε, ένα σύστημα διαχείρισης. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό. Χαβιέ ε, Λόπες. Ο Χαβιέ Λόπες. Σας ευχαριστώ πολύ. Διάβασα και διαβάζω την μελέτη αυτή με μεγάλη προσοχή. Η έκθεση αυτή αναλύει τις συγκεκριμένες ανάγκες των μικροεπιχειρήσεων και των μικροεπιχειρηματιών και τα, ε, τις, ε, τις χρηματοπιστωτικές λύσεις που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Microfinance Facility, 27 προγράμματα με 5 χώρες. Ε, πρέπει να μελετήσουμε καλά τις πληροφορίες που μας δώσατε και θέλαμε να ε, μιλήσουμε για κάποια από τα συμπεράσματα τα οποία αναφέρεται εδώ. Καταρχήν λέτε ότι δεν υπάρχουν ε, προηγούμενες μελέτες όσον αφορά τις ανάγκες ε, που εκφράζουν οι πιθανοί δικαιούχοι, όπως ας πούμε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θα ήθελα να γνωρίζω ποιες συνέπειες έχει κάτι τέτοιο και πώς θα μπορούσε να ρυθμιστεί. Στην περίπτωση του Κοινωνικού Ταμείου υπάρχουν συγκεκριμένες στρατηγικές επενδύσεις για αυτές τις εταιρείες, μικροεπιχειρήσεις και θέλαμε να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις ε, με μια συγκεκριμένη πολιτική ε, για την ε, υλοποίηση ή την κατάργηση ορισμένων από αυτά τα προγράμματα. Επίσης, την δημιουργία ιδιωτικού κεφαλαίου που επικρίνεται, αλλά και άλλους μηχανισμούς, το European Progress Microfinance Facility, που έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει ιδιωτικό κεφάλαιο και έχει και πολλές ε, δυνατότητες ε, ε Μια τελευταία παρατήρηση για την δυσκολία που υπάρχει ως προς την ανάγνωση του κοινωνικού αντικτύπου που έχουν αυτές οι μικροπιστώσεις. Στην Επιτροπή μιλούσαμε για το θέμα αυτό. Το κοινωνικό αντίκτυπο, τον κοινοοικονομικό αντίκτυπο που έχει η μικροπίστωση και θυμίζει η έκθεση ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες επαρκής για το προφίλ των ε, ε, δικαιούχων, την επιβίωση των έργων, το κέρδος αυτών των ανθρώπων, δηλαδή ποιος είναι ο πραγματικός καμένος Δεν είναι εύκολο δηλαδή να αναγνώσουμε σωστά όλα τα εργαλεία. Πρέπει όλοι να σκεφτούμε ότι πρέπει να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για να μπορέσουμε να παράσχουμε και εμείς επαρκής, επαρκή ενημέρωση και να έχουμε μια σωστή εικόνα. Κύριε Μάκιντάιρ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα την έκθεση. Και πολύ χαίρομαι που σας ξαναβλέπω εδώ επίσης, γιατί πιστεύω πως ε, το να καταλάβει κανείς ε, την αποτελεσματικότητα των ε, προγράμματων και του τρόπου με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ βασικό για να ξέρουμε ότι έχει προστιθέμενη αξία αυτό που κάνουμε. Δηλαδή ε, να ξέρουμε ότι όντως ε, επιτύχαμε αυτό που είχαμε στόχο ως νομοθέτες. Είναι ωστόσο κάπως ανησυχητικό ότι βρήκατε τέτοιες αδυναμίες στον προγραμματισμό και το σχεδιασμό της στήριξης. Είμαι ευτυχής που τις βρήκατε βέβαια αλλά ε, αυτό που εσείς ιδιαίτερα τονίσατε ήταν ότι δεν υπάρχει ουσιαστική και πλήρης ανάλυση των αναγκών. Διορθώστε με αν ε, ε, κάνω λάθος. Πάντως έχω την εντύπωση ότι στην ουσία πετάμε χρήματα στο πρόβλημα, χωρίς όμως να έχουμε αξιολογήσει ακριβώς τι χρειάζεται και από τις διάφορες σας συστάσεις ε, προκύπτει αυτό. Η πρώτη σας σύσταση είναι ότι τα κρατημέλη θα πρέπει διαρκώς να προβαίνουν σε αναλύσεις αναγκών. Κατά κάποιο τρόπο είναι θα να έχουμε κάνει το αντίθετο από το κανονικό. Ότι δηλαδή πρέπει κανονικά να έχουμε κάνει μια σωστή αξιολόγηση των αναγκών πριν αποφασίσουμε να δαπανίσουμε χρήματα. Αυτό είναι σημαντικό μήνυμα. Τα χρηματοπιστωτικά στα μέσα θα έπρεπε να προσφέρονται υπό τον όρο ότι τα κράτη-μέλη έχουν ένα στιβαρό ε, σύστημα διαχείρισης κινδύνου. Αυτό το στηρίζω. Κατά κάποιο τρόπο με εντυπωσιάζει κιόλα που δεν υπάρχει ήδη ένα τέτοιο μηχανισμό. Πολύ θα ήθελα να ακούσω το σχολείο σα σχετικά. Και τέλο, η σύσταση παρθμών 3 ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα φτάσουμε στους ανέργους και στους ευάλωτους ανθρώπους. Είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που δημιουργούν οι ίδιοι την ε, δική τους δουλειά. Να εξετάσουμε δηλαδή τους ανέργους και να σχεδιάσουμε τα μέσα στήριξης με τρόπο ώστε να βοηθήσουμε μικροεπιχειρηματίες που έχουν ιδέες και είναι πρόθυμοι και ικανοί να δημιουργήσουν την ίδια τους θέση εργασίας και έτσι να βγουν από τις λίστες των ανέργων. Πολύ σημαντικό λοιπόν είναι να στοχεύσουμε ακριβώς αυτού στους ανθρώπους. Και όλα αυτά βέβαια συνδέονται στενά με την αξιολόγηση και την κατανόηση των αναγκών. Αυτά τα σχόλιά μου και ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρία Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν είναι υπέρ κατά το ότι συζητήσαμε την έκθεση αυτή στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού αρχέ τη εβδομάδα, αλλά βλέπω, είναι ενδιαφέρον να βλέπει κανεί την ίδια έκθεση και από τι δύο πλευρέ, γιατί ακού άλλα πράγματα από του συναδέλφου. Θέλω να τονίσω, ήδη τα ανέφερα κάποια από αυτά και στην άλλη επιτροπή. Προφανώς η οικονομική υποστήριξη είναι σημαντικό θέμα και μπορούμε να το συζητήσουμε σήμερα από μια άποψη τεχνικής απασχόλησης. Έχω επιφύλαξη αν ξέρουμε ποιες είναι οι ανάγκες των μικροεπιχειρηματιών, διότι η έκθεση αναφέρει κάποιες από τις ανάγκες αυτές, όχι όμως όλες. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι λοιπόν ότι εντοπίσαμε τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρηματιών και την σωστή, ε, το σωστό εντοπισμό των αναγκών αυτών που είναι απαραίτητη προϋπόθεση σωστή χρήση των ευρωπαϊκών πόρων. Δεν πειράζει δηλαδή αν είναι εργαλεία ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου ή όχι. Φαίνεται επίσης ότι συγκρίνουμε άσχετα πράγματα σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά εγώ το θέμα το βλέπω λίγο πιο ε, οπτικά. Οι στόχοι των χρηματοδοτικών εργαλείων είναι τελικά οι ίδιοι. Η, μικρο, η παρουσίαση μη, μικροπιστώσεων, η ενίσχυση των μικροπιστώσεων και οι συνέργειες μεταξύ τους, διότι πρέπει να βρούμε μια συνέργεια μεταξύ των διαφορετικών αυτών εργαλείων, το αποτέλεσμα δε των συνεργειών θα είναι αυτό, μάλλον και το αποτέλεσμα είναι αυτό που πρέπει να δούμε. Κάτι άλλο που προσπαθούσα να εξηγήσω τη Δευτέρα στο δικαστήριο είναι ότι δεν έχω πληροφορίες για την βιωσιμότητα των μικροεπιχειρήσεων μετά από μία συγκεκριμένη περίοδο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Αν αυτοί, αυτές οι επιχειρήσεις ε, είναι κερδοφόρες, βιώσιμες, αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να προσθέσω στους δείκτες. Τελευταία παρατήρηση. Ivanova personally was uh, listening Uh, yesterday at about budget. Κάτι που δεν άκουσα είναι αυτό που το είπε η κυρία Ιβάνοβα. Το budget based performance ε, παραδείγματα. Στην έκθεση δεν υπάρχουν καλά παραδείγματα, καλές πρακτικές που θα βοηθούσαν μια περαιτέρω αξιολόγηση των έργων. Και η ανακοίνωση πρέπει να αλλάξει για την χρηματοδότηση Τελευταίο θέμα, το δεν ξέρω αν αυτό είναι ερώτημα προς το, δικαστήριο, την Κομισιό, προς το ελεγκτικό συνέδριο την Κομισιόν. Τα οικονομικά εργαλεία στον τομέα του κοινωνικού ταμείου είναι δύσκολο εγχείρημα. Βρήκατε ωστόσο τους βασικούς λόγους που οι πόροι αυτοί έχουν χαμηλή μόχλευση. γιατί αυτό είναι αυτό που θα εξετάσω αρκετά στην έκθεσή μου για την απαλλαγή του 2014. Υπάρχουν κάποιες ιδέες από πλευρά σας. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις. Ελπίζω να μπορείτε να απαντήσετε. The good answers to them. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές για τις ε, πολύ ε, σωστές ερωτήσεις και παρατηρήσεις σας. Ε. Οι επιχειρηματίες της Ευρώπης, οι είναι πολύ σημαντικοί διότι εκπροσωπούν το 90% στην Ευρώπη και δεδομένου του αριθμού των επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μικροεπιχειρήσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ ε, σωστές οι ερωτήσεις αυτές. Θα ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση. Είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς ε, πολύ συγκεκριμένα θετικά πράγματα στην εκθεσία, αυτή. Αν όμως υπάρχει κάτι θετικό, θα έλεγα ότι με βάση τα προγράμματα που επισκεφτήκαμε θα έλεγα ότι το πιθανότερο είναι να καταφέραμε να φτάσουμε τους μικροεπιχειρηματίες της Ένωσης. Το θέμα από εκεί πέρα είναι πόσο αποτελεσματική ήταν αυτή η προσπάθεια, αλλά ε, νομίζω ότι πράγματι φτάσαμε σε αυτούς τους βρήκαμε, του εντοπίσαμε. Το θέμα είναι αν αυτό έγινε με τρόπο ε, οικονομικά αποδοτικό, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω και πιο συγκεκριμένα σε ερωτήσεις σας. Κύριε Σούλσε, αναφέρατε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο τέθηκε και τη Δευτέρα στην ε, ε, Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ε, ρωτήσατε μήπως ε, συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια ε, συγκρίνοντας τα δύο ταμεία. Καταλαβαίνω την ανησυχία σας. ε, τίθεται το ερώτημα εάν το ένα μέσο είναι καλύτερο από το άλλο, αλλά όχι, δεν είναι αυτό το θέμα, δεν προσπαθούμε να τα συγκρίνουμε. Προσπαθήσαμε πιο πολύ να αναλύσουμε ανεξάρτητα το καθένα από αυτά, διότι όπως ανέφερε η κυρία Τραπολόβα, και τα δύο αποτελούν πηγή χρηματοδότησης για τους μικροεπιχειρηματίες μας παρότι υπάρχουν κάποιες διαφορές στους στόχους των δύο ταμείων. Έχουν τον ίδιο στόχο να βελτιώσουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικροεπιχειρήσεων και από τη φύση τους έχουν κάποιες ομοιότητες, ε, έχουν κάποια κοινά όσον αφορά τη δομή τους ε, ε, όσον αφορά τους όρους, χρήσης ε, των πόρων, αλλά τελικά εναπόκειται ε, στο εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο να επιλέξει το πιο κατάλληλο μέσο για την κάθε περίπτωση. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, μπορεί να είναι πιο χρήσιμη μια χορηγία, σε άλλες περιπτώσεις μια πίστοση, σε, στην τρίτη περίπτωση ένα από τα οικονομικά μέσα του ESF. Ίσως ε, λοιπόν ε, και μόνο από πλευράς κόστους μπορεί να δίδεται η εντύπωση ότι προσπαθούμε να συγκρίνουμε τα διάφορα ταμεία, αλλά το κάθε ταμείο εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό και προσπαθούμε με την έκθεση αυτή να δώσουμε μία πιο πλήρη εικόνα, ώστε όταν λαμβάνονται οι αποφάσεις αυτές να λαμβάνονται ε, πιο εμπεριστατωμένα θέσατε και το θέμα της επιλογής των κρατών μελών. Είναι ειδική η έκθεση αυτή. Σε άλλες τέτοιες ειδικέ εκθέσεις εξετάζουμε 4, 5, 6 κράτη-μέλη. Στις περιπτώσεις αυτές επιλέξαμε τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την, και τη Ρουμανία. Την Πολωνία και τη Ρουμανία. Γιατί, διότι η Πολωνία, η Γέρμανη και η Ιταλία έχουν τις μεγαλύτερες πιστώσεις για την υποστήριξη των ε, νεοφιών επιχειρήσεων και αντιπροσωπεύουν το 75% των συνολικών πόρων. Από την άλλη, η Ρουμανία και η Ισπανία δεν ε, ε, έχουν διαθέσει πολλά χρήματα σε αυτούς τους κωδικούς. Η Ρουμανία είναι από τους μεγαλύτερους δικαιούχους όμως του EPMF. Προσπαθούμε λοιπόν πάντα να δίνουμε ισορροπημένη εικόνα των μεγαλύτερων δικαιούχων και γεωγραφικής κατανομής, ώστε ο λογιστικός έλεγχος ε, να δίνει μια καλή επισκόπηση. Και πέρα από αυτές τις επισκέψεις στα κράτη-μέλη, κάναμε και μια έρευνα 18 διαχειριστικών αρχών ε, σε 14 κράτη-μέλη που είναι αρμόδια για 22 επιχειρησιακά προγράμματα του ESF. Και νομίζω ότι γενικά είμαστε ικανοποιημένοι με την ανταπόκριση που ανέρχεται ε, σχεδόν σε 90% και έτσι συλλέξαμε πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες τους για την παροχή χρηματοδότησης σε μικροεπιχειρηματίες. Αναφέρθηκε αρκετές φορές η αξιολόγηση. Πράγματι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, διότι αν ξεκινήσουμε από λάθος σχεδιασμό, τότε μάλλον θα καταλήξουμε και σε λάθος κατεύθυνση. Γι' αυτό, για να πετύχουμε καλά αποτελέσματα, θα πρέπει να έχουμε σωστό σχεδιασμό και σωστή εφαρμογή. Γι' αυτό βρήκαμε ότι η αξιολόγηση ήταν σημαντική έλλειψη στο όλο εγχείρημα και βέβαια είναι πολύ σημαντικό και το ποσοστό επιβίωσης ε, για την βιωσιμότητα των προγραμμάτων. Είναι ένας από τους σημαντικότερους δείκτες απόδοσης που αποδεικνύει ε, αν ήταν επιτυχές το πρόγραμμα. Δηλαδή αν ε, επιβιώσει μόνο για ε, ένα-δύο χρόνια ή αν δεν επιβιώσει καθόλου τότε ίσως να μην άξει τον κόπο για επένδυση σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Όλα αυτά σχετίζονται με αυτά που ανέφερε η κυρία Μάκιντάιερ σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, διότι στο κάτω-κάτω το θέμα που τίθεται είναι όχι μόνο εάν δαπανίσαμε τα χρήματα, αλλά εάν τα δαπανίσαμε για να πετύχουμε καλά αποτελέσματα και να βελτιώσουμε την ζωή των πολιτών μας. Ε, και έτσι επανερχόμαστε στην ε, αξιολόγηση των αναγκών. Η Κομισιόν έχει αποδεχτεί όλες τις συστάσεις εκτό από την τελευταία, αλλά νομίζω ότι ακόμα και εκεί η σύσταση να αξιολογηθεί το κόστος για τα διάφορα μέσα βασίζεται στην καλή πρακτική που ήδη έχει εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτείνουμε λοιπόν επικαιροποίηση των πληροφοριών αυτών, διότι Πιστεύουμε ότι το μοίρασμα των βέλτιστων πρακτικών ε, μπορεί να αποτελέσει προστιθέμενη αξία για τους δικαιούχους. Και ε, επίσης ε, έχουμε αυτό που ανέφερε η κυρία Τραπαϊόβα. Εάν γνωρίζουμε το κόστος μπορούμε να ζητήσουμε καλύτερους τρόπους να ε, πετύχουμε την προστιθεμένη αξία. Προσπαθώ να βρω συγκεκριμένα παραδείγματα για να απαντήσω στην κυρία Ντελαμπαγιώβα. Νομίζω ότι στην σελίδα 15 στο σχήμα 2 βλέπουμε ένα καλό παράδειγμα σε αυτή την αξιολόγηση αναγκών που πραγματοποιήθηκε ε, εξετάζοντας ε, τις ανάγκες των νεοφυών επιχειρήσεων. Η μελέτη αυτή βασίστηκε σε ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση της μικροχρηματοδότησης. Μπορεί τα αποτελέσματα να μην είναι αυτά που θα περιμένατε, αλλά άλλο καλό παράδειγμα που σχετίζεται με τη συζήτηση σχετικά με το κόστος εφαρμογής είναι η μελέτη της Κομισιόν του 2011, όπου εξετάζει την ε, εφαρμογή αυτών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Πιστεύουμε ότι έτσι παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες ε, για αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις, ε, κάτι που οδηγεί σε πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων. Θα χαιρόμουν ακόμα περισσότερα, αν θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα περισσότερα καλά παραδείγματα, αλλά αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει. Από προηγούμενες εκθέσεις όμως που έχουμε συζητήσει γνωρίζετε ότι προσπαθούμε να μην δίνουμε μία, ε, μία μονομερή ανισορροπή εικόνα. προσπαθούμε να εξετάζουμε και τις ευέλτιστες πρακτικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Διαμπάλοβα. Ναι, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, διότι αυτή τη στιγμή είμαστε μόνο τέσσερις Ευρωβουλευτέ, πέντε ευρωβουλευτέ από τέσσερις πολιτικές ομάδες. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Και ω Αντιπρόεδρος τη ε, Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού, θα ήθελα να πω ότι δεν συνηθίζεται οι εκπρόσωποι του Ελεκτικού Συνεδρίου να επισκέπτονται τις τεχνικές επιτροπές. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την κυρία Ιβάνοβα, διότι είναι πολύ χρήσιμη αυτή η επίσκεψη, αυτή η επίσκεψη και ως ε, μέλος ε, της Επιτροπής ε, Κοντ, ε, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ χρήσιμο για μας, διότι χρειαζόμαστε αυτές τις τεχνικές και συγκεκριμένε πληροφορίες. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω και να προτείνω να το κάνουμε αυτό πιο συχνά, διότι έχουμε πολλές ειδικέ εκθέσεις, ειδικέ συζητήσεις, έχουμε ακροάσεις για την απαλλαγή για το 2014. Ίσως αυτή θα ήταν μια ευκαιρία να παρευρεθείτε ώστε να είσαστε παρούσα όταν συζητάμε την, ε, για το πώς δαπανώνται τα ευρωπαϊκά χρήματα στον τομέα της απασχόλησης. Ευχαριστώ και ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που το οργανώσατε αυτό. Η κυρία Ιβάνοβα, σας ευχαριστώ πολύ διότι είναι πολύ χρήσιμη αυτή η πληροφορία για μας και θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία και πάλι να, διαφημίσω, να την επικείμενη έκθεσή μας ε, διότι είναι ένα θέμα που σας ενδιαφέρει και σας. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι πολύ σύντομα θα δημοσιεύσουμε την ε, εκθεσή μας ε, για τις ομάδες της δράσης για τους νέους και θα εξετάσουμε την εφαρμογή της εγγύησης των νέων σε επίπεδο κρατών μελών. Όποτε με προσκαλείτε έρχομαι με πολύ χαρά και σας ευχαριστώ για την εξαιρετική συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Σας καλούμε τώρα λοιπόν να μας παρουσιάσετε την έκθεση που αναφέρατε. Πολύ θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε τι έχετε να πείτε για την έκθεση αυτή. Επίσης θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Εμείς ε, Καταρχά θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Ελεκτικό Συνέδριο για, τον για την επαγγελματική προσέγγιση και σε αυτή την ακρόαση και στις άλλες. Μας βάζετε πολλές δουλειές, το είχα πει και στην κυρία Ιβάνοβα, αλλά νομίζουμε ότι η έκβαση των συζητήσεων είναι εξαιρετικά χρήσιμες για να μπορούμε να παίρνουμε σωστές αποφάσεις στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το ελεκτικό συνέδριο. Για τη συγκεκριμένη έκθεση θέλω να τονίσω ένα θέμα που δεν αναφέρθηκε. Το follow-up στις συστάσεις του συνεδρίου. Ιδίως τις τρεις συστάσεις που εντόπισαν πιθανότητες βελτιώσεων για στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται τα εργαλεία αυτά κυρίως στο κοινωνικό ταμείο. Και τονίζω ότι το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την περίοδο 14-20 που δεν έχει δει ακόμα το, συνέδριο διότι εξετάζει την εφαρμογή ακόμα του πλαισίου 2013. Το νέο πλαίσιο λοιπόν βελτιώνει της, ε, της διαδικασίας στη στο θέμα των υποχρεώσεων των κρατών μελών και των, ε, τα, τις δυνατότητες που έχουν οι δικαιούχοι για να αντιμετωπίσουν τις ε, συστάσεις και τα ευρήματα του ελεγκτικού συνεδρίου. Να πω λοιπόν και εγώ ότι πολύ στα ευρήματα του συνεδρίου δεν μας εκπλήσουν και πολύ τουλάχιστον διότι πολλές από τις αδυναμίες που παρατηρήσαμε όταν αναλύαμε την εμπειρία με το προηγούμενο πλαίσιο και τα χρηματοδοτικά μέσα που εμπεριέχει το τελευταίο, όταν κάναμε τη δουλειά μας την ε, πρόταση βελτίωσης του νέου κανονιστικού πελεσίου, εμείς πιστεύουμε πραγματικά ότι εμείς όντας εδώ το, ότι αν είμαστε εδώ το 2022 θα μπορέσουμε να ακούσουμε ακόμα πιο θετικά μηνύματα από πλευράς ελεκτικού συνεδρίου για την, αξιοποίηση, για την αξιολόγηση του πώς μπορεί περαιτέρω να βελτιωθεί ο τρόπος ε, χρήσης ε, των ε, όλων των χρηματοδοτικών μέσων, ιδίω δε του κοινωνικού ταμείου και το πώς λειτουργούν. Μια τελευταία απάντηση στο ερώτημα της κυρίας Λαμπάγιοβα για το βαθμό μόχλευσης. Όντω, ε, σωστά το λέτε ε, το ελεκτικό συνέδριο ότι υπάρχουν διαφορετικές ε, διαφορετικά επίπεδα μόχλευσης σαν χρηματοδοτικό μέσο, χαμηλότερο για το κοινωνικό ταμείο, αλλά ένας μόνο παράγοντας που μπορεί κάλλιστα να το εξηγήσει αυτή τη μειωμένη, αυτό το μειωμένο ποσοστό μόχλευσης στο κοινωνικό ταμείο είναι ο στόχος της χρήσης ε, του εργαλείου αυτού να χρησιμοποιηθεί δηλαδή η μικροψη πίστοση για να βοηθήσει τους πλέον ευάλωτους στην Ένωση αφενός και να δημιουργήσει μία αγορά για τέτοια πίστοση, για τέτοια ε, για τέτοιο αμορφιδανισμό που είναι ακόμα κάπως περιορισμένος. Μην ξεχνάτε ότι η αγορά δεν είναι ανεπτυγμένη αρκετά και άρα λιγότερο ελκυστική για το ιδιωτικό κεφάλαιο που εξηγεί το χαμηλότερο επίπεδο των μέσων αυτών. Ωστόσο, εμείς πιστεύουμε και το επιβεβαίωσε αυτό το ελεκτικό συνέδριο ότι η χρήση αυτής, αυτών των μέσων για την υποστήριξη των ευάλωτων ατόμων έχει πλεονεκτήματα και παρά το χαμηλό επίπεδο ε, των επιπτώσεων συνεχίζεται για άλλους λόγους. Προφανώς ωστόσο η χρησιμοποίηση των οικονομικών μέσων δεν είναι πανάκια στην συγκεκριμένη περίπτωση και ίσως σε μερικές περιπτώσεις να είναι πιο χρήσιμη η δωρεάν, ε, ο δανεισμός, ε, η δωρεά. Θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Σας όλους. Αυτά είναι τα ερωτήματα που έχουμε να απαντήσουμε όταν συναντάμε τους ψηφοφόρους μας. Πού πάνε τα λεφτά, τι τα κάνετε τα λεφτά, ποιο είναι το αποτέλεσμα των αποφάσεων που λαμβάνετε για τα χρήματα. Και έτσι είναι ακόμα πιο σημαντικό για μας να σας καλούμε κάθε φορά. Με την επόμενη ευκαιρία λοιπόν, όταν θα έχετε να μας πείτε πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα. Ελπίζουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα και έτσι να μπορούμε να δώσουμε αυτό το ευχάριστο μήνυμα προς τους ψηφοφόρους μας, αυτό που είναι το πιο σημαντικό. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε και ευχαριστώ και στην Επιτροπή. Αυτό σημαίνει τώρα ότι εδώ ολοκληρώθηκε αυτή η συνεδρίαση. Αρχίσαμε στις 9 το πρωί σήμερα και θα τα ξαναπούμε στις 12 Οκτωβρίου και στις 13 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ όλους. Καλό σας απόγευμα.